Diamo inizio. Benvenuti a tutti. Ας ξεκινήσουμε. Καλωσορίσατε όλοι. Ξεκινάει η συνεδρίαση της Επιτροπής. Καταρχήν, όπως βλέπετε, να είμαι, εδώ είμαι. Ε, δεν ε, θα πάω να γίνω υπουργό Γεωργία ε, στη χώρα μου. Ευχαριστώ συνάδελφοι για τα mail που μου στείλατε, αλλά δεν θα πάω. Ξεκινάμε λοιπόν την σημερινή συνεδρίαση. Εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Να σας πω ότι έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες της Επιτροπής μας. να εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 4ης Μαρτίου, 10ης Μαρτίου, 18ης και 19ης Μαρτίου και 25ης Μαρτίου. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, πριν από το πέρας της συνεδρίασης, τα πρακτικά αυτά θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Να σας πω επίσης ότι η σημερινή συνεδρία αναμεταδίδεται στο ίντερνετ. Και τώρα περνάμε στην ε, δημόσια κρόση όσον αφορά τις εμπειρίες των νέων κρατών μελών στην εφαρμογή της κοινή γεωργικής πολιτικής από το 2009 στο 2013. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να καλωσορίσουμε έξι εμπειρογνώμονες που θα μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους για τις εμπειρίες των ε, κρατών μελών τους μετά από την εφαρμογή της κοινή γεωρικής πολιτικής. Είναι σκόπιμο να σημειώσουμε ότι η εμπειρία εφαρμογής είναι σημαντική για να επιτευχθεί ο στόχος της απλοποίησης που έχουμε θέσει στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Θα υπάρξουν λοιπόν τρεις, ε, τρία τμήματα με δύο εμπειρογνώμονες ανά τμήμα και κάθε φορά θα ακολουθεί συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής μας. Τρία τμήματα λοιπόν συζήτησης, αφού θα έχουμε ακούσει κάθε φορά δύο εμπειρογνώμονες, θα γίνεται συζήτηση με τους συναδέλφους που θα θελήσουν να πάρουν τον λόγο, ακόμα δύο και τα λοιπά και τα Πρώτο τμήμα λοιπόν αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και τα καθεστώτα ενιαίας στρεματικής ενίσχυσης. και σε στα ελληνικά. Ναι, τα αρχικά. Πρώτος ε, εμπειρογνώμονας είναι ο κύριος Βόιτσεκ Πομάιντα, που είναι διευθυντής του Ιδρύματος Προγραμμάτων Παροχής Βοήθειας για τη Γεωργία και τέος διευθυντής του αντίστοιχου Πολωνικού Οργανισμού Πληρωμών. Θα μας μιλήσει για την εμπειρία της Πολωνίας στην εφαρμογή της κοινή γεωργικής πολιτικής από τα πρώτα έτη της ως μέλος της Ένωσης. Επόμενος ομιλητής αυτού του πρώτου τμήματος θα είναι ο κύριος Μπάλας Γιόρφη, που είναι πρόεδρος του Ουγγρικού Γεωργικού Επιμελητηρίου και θα μιλήσει σχετικά με τις προσδοκίες των αγροτών της, Γεωργ... της Ουγγαρίας από τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής βάσει των εμπειριών που είχαν ε, από τη μέχρι του δεφαρμογή της. Ε, Καλώ τους εμπειρογνώμονες να πάρουν το λόγο για 10 λεπτά maximum ο καθένας. Παρακαλώ. Ο κύριος Πομάιντα. Θέλω, this, want Θέλει ο κύριος Δέσης λόγο πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έγινε μια παρατήρηση για το σχηματισμό κυβέρνησης στην Ιταλία θα έλεγα ότι εμένα θα με ανησυχούσε ιδιαίτερα το να δεχθεί, εάν δεχόταν, ο πρόεδρος της Επιτροπής μας ε, υπουργικό θόκο στην Ιταλία και να χωρούσε για Ρώμη ε, σε μια περίοδο που εδώ έχουμε να κάνουμε τόσο σημαντικές ε, μεταρρυθμίσεις και σοβαρές αποφάσεις. Θα πρέπει, πιστεύω, ο πρόεδρος της Επιτροπής μας να παραμείνει εφό ετάχθη μέχρι το τέλος της τουλάχιστον. Ο κύριος Πομάιντα, λοιπόν, ο πρώτος μας εμπειρογνώμων για 10 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα και το θεωρώ και τιμή μου που μπορώ να συμμετάσχω στη συνεδρία σε αυτή της Επιτροπής σας. Είναι μεγάλη και σημαντική ευκαιρία για μένα να μπορώ μαζί σας να ανταλλάξω απόψεις όσον αφορά την εφαρμογή της κοινή γεωργικής πολιτικής της χώρας μέλη. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τις πληρωμές τους οργανισμούς πληρωμών και τις εμπειρίες που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα. Εγώ συμμετέχω σε έναν από αυτούς τους οργανισμούς. Καταρχήν από το 2003 μέχρι το 2005 συμμετείχα τότε που έγινε και η προσχώρηση της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε ασχολήθηκα με τις πρώτες πληρωμές που πήγαν στην Πολωνία εκείνη την εποχή. Όπως γνωρίζετε, η εμπειρία μας είναι ίδια με την εμπειρία που έχουν και άλλες χώρες οι οποίες προσχώρησαν εκείνη την εποχή μαζί με την Πολωνία δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την αρχή υπήρχαν πολύ συγκεκριμένοι στόχοι. Τι σήμαιναν αυτοί για τα κράτη-μέλη. Εδώ φυσικά θα επικεντρωθώ στην Πολωνία, τη δικιά μου τη χώρα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν έπρεπε να ε, προχωρήσουμε σε κάποιες προσαρμογές του νομικού μας συστήματος, και των ρυθμίσεών μας και κατά την προενταξιακή περίοδο, αλλά και μετά την ένταξη της Πολωνίας. Έπρεπε να εφαρμόσουμε και εμείς το νέο κοινοτικό κεκτημένο, αλλά έπρεπε να ετοιμάσουμε και τους θεσμούς της χώρας να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κεκτημένου αυτού. Άρα λοιπόν χρειάστηκε πολλή δουλειά, η οποία μας επέτρεψε τελικά να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τις αγορές μας, να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στις κοινοτικέ αγορές και μας έδωσε και κίνητρα να δουλέψουμε και να ανταγωνιστούμε τελικά με τους ε, εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μερικές φορές ήταν πολύ πιο ισχυροί από μας. Τώρα την περίοδο 2004 με 2012 η Πολωνική Γεωργία πήρε χρήματα συνολικά 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ συμπεριλαμβάνουμε και το εθνικούς και τους κοινοτικούς προπολογισμούς, τα κονδύλια δηλαδή και τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά. Βέβαια, ήδη τότε συνεισφέραμε και εμείς τον ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Έπειτα, εδώ βλέπετε το πρώτο και το δεύτερο πυλώνα και τι έχουμε δώσει. Αν ψάξετε εδώ στη γραμμή να βρείτε την Πολωνία, θα δείτε ότι εμείς βρισκόμαστε στο επίπεδο των 320. Ανεκτάριο. Κάτω από το μεσόρο, δηλαδή, που είναι 445 για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή των 27. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Τώρα, γιατί η Πολωνία αποφάσισε να συμφωνήσει με το καθεστώς ε, ενιαίων ενισχύσεων. Αυτό έγινε και ακόμα στα πλαίσια του ΠΟΕ είναι κάτι το οποίο θεωρείται αποσυνδεδεμένο από την παραγωγή. Και η εμπειρία μας από το 2005 μας έδειξε ότι ένα απλοποιημένο σύστημα θα είχε περισσότερες πιθανότητες να υιοθετηθεί και από τις 15 παλιές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα λοιπόν μας επέτρεψε να απορροφήσουμε τα κονδύλια τα οποία προορίζονταν τα πρώτα χρόνια για την πολωνική γεωργία και έγιναν απλοποίησεις και από τους γεωργούς αλλά και για τους γεωργούς. Πιο απλοποιημένες δηλαδή διαδικασίες προκειμένου να συμπληρώσουν τις αιτήσει τους ή προκειμένου να μπορούν να τις διορθώσουν εφόσον χρειάζεται αυτό. Γιατί τώρα ήταν τόσο σημαντική για την Πολωνία η απλοποίηση, διότι η Πολωνία, μιλάμε για 312.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε, με πάνω από 34 εκατομμύρια ε, έκταση για τις γεωργικές ε, εκτάσεις και έπειτα υπάρχει και 45% είναι το ποσοστό σε σχέση με τη χώρα μας ολόκληρη. 2 εκατομμύρια είναι οι καταγεγραμμένοι με ένα μέσο όρο 10,38 εκτάρια. Το 2000 Ίσως η αύξηση να μην ήταν πολύ σημαντική, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι από τότε και μετά αυξήθηκε πάρα πολύ και σήμερα είναι 10,30 το εκτάρια. Εδώ έχετε το μέσο όρο επίσης 1,4 εκατομμύρια αιτήσει για ε, το, τις ενισχύσεις αυτές. Μπορείτε βέβαια να συγκρίνετε με το τι γίνεται στις δικές σας τις χώρες, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας κάθε φορά πόσοι είναι οι αγρότες σε κάθε χώρα. Επιπλέον, στην Πολωνία έχουμε κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσει για το καθεστώς ενιαίων ενισχύσεων. Ανά εκτάριο έχουμε πολύ βασικές και γεωργικές προϋποθέσεις αλλά και περιβαλλοντικές. Οι πληρωμές αναεκτάριο καθορίζεται και λαμβάνεται υπόψη και η περιοχή αλλά και το προϊόν πρέπει να είναι επιλεγμένο. Υπάρχουν ε, προϊόντα από περιοχές οι οποίες θεωρούνται κατά από καλές συνθήκες περιβαλλοντικά και είναι κάτι το οποίο φυσικά επαληθεύουμε. Αν υπάρχει και η πολλαπλή και όλες οι άλλες οι προϋποθέσεις που θέλουμε. Και υπάρχει και μία περίοδος σταδιακής μείωσης. Τώρα εδώ η επόμενη διαφάνεια σας δείχνει 2004 με 2013 την περίοδο αυτή. Βέβαια Ακόμα είμαστε στα μέσα του 2013 και οι πληρωμές για το 2013 δεν έχουν γίνει ακόμα. Αλλά βλέπετε στον πίνακα αυτό τα ποσοστά. Σε τι επίπεδο ποσοστών βρισκόμαστε δηλαδή όταν μιλάμε για ευρωπαϊκές ε, πληρωμές. Σε πράσινο και σε μπλε βλέπετε τα χρήματα τα οποία παίρνουμε από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Βέβαια υπάρχει και ο αλγόριθμος, ο μηχανισμός εκείνος τον οποίο διαπραγματευτήκαμε πριν προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσχυε τα πρώτα χρόνια μέχρι το 2006, ότι δηλαδή ένα μέρος των κονδυλίων μεταφέρονταν από την περιφερειακή ανάπτυξη στις άμεσες ενισχύσεις. Εδώ είναι δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Ξεκινάμε βέβαια με την περίοδο 2004 με 2006 και εδώ είναι περίπου 5 ε, δισεκατομμύρια ευρώ και μετά βλέπετε και τις επόμενες χρονιές τι έγινε με τις πληρωμές και βλέπετε εδώ πως αλλάζουν τα ποσά και η κατανομή. 3,3 δις περίπου το χρόνο. Κοιτάξτε και την τελευταία κολόνα για το 2012. Δεν είναι βέβαια πλήρης γιατί οι πληρωμές ακόμα δεν έχουν γίνει όλες. Ποια είναι τώρα τα πλεονεκτήματα του ενιαίου καθεστώτος ενισχύσεων. Για μας το σύστημα αυτό ανταποκρίνεται στα μέτρα στήριξης τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πληρωμή δηλαδή έτσι συνδέεται με τις προϋποθέσεις για μια συγκεκριμένη περιοχή. Είναι κάτι το οποίο επίση μας βοηθάει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και τα κονδύλια τα οποία φτάνουν σε εμά τους αγρότες. Διότι υπάρχει ανάλυση ανά εκτάριο. Μας επιτρέπει επίσης να αποφύγουμε το πρόβλημα των κονδυλίων τα οποία τελικά δεν απορροφούνται. Η χρήση του συστήματος αυτού μας βοηθάει να μειώσουμε και το κοινωνικό κόστος. Και θέλω εδώ να αναφερθώ και στις αλλαγές. Μία αλλαγή στο σύστημα δεν νομίζω ότι θα γινόταν ευπρόσδεκτη στους ε, αγρότες οι οποίοι δεν θα έχουν εμπιστοσύνη. Θα φοβούνται ότι δεν θα βελτιωθεί η κατάστασή τους με τις αλλαγές αυτές μια τέτοια αλλαγή μάλλον θα κόστιζε περισσότερο για να μπορέσει και να εφαρμοστεί και σίγουρα θα χρειαζόταν καιρός για να γίνει η προσαρμογή αυτή και θα αυξανόταν και το ε, διοικητικό κόστος. Τώρα το σύστημα αυτό του καθεστώτος ενίων ενισχύσεων δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κάποιο άλλο σύστημα, για παράδειγμα το σύστημα πληρωμών σε νέους ε, αγρότες ή κονδύλια που έχουν να κάνουν με την παραγωγή. Και για να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα, θέλω να αναφερθώ εδώ στο κόστος στην Πολωνία σε σχέση με τις υπηρεσίες, αν μπορώ να πω, των άμεσων ενισχύσεων. Το ετήσιο κόστος είναι 100 ευρώ για την επεξεργασία μίας αίτησης. Τον ΟΚΕ συνολικά 140 εκατομμύρια. Κάτι το οποίο περιλαμβάνει τις επιθεωρήσεις επιτόπου, το σύστημα ταυτοποίησης. Αν δείτε λοιπόν την ανάλυση ανά χρόνο και λάβετε υπόψη σας το συνολικό ποσό που πληρώνεται σε κάθε χώρα, τελικά καταλήγουμε σε ένα 4,5% διοικητικό κόστος. Τώρα ποιες είναι οι προσδοκίες για το μέλλον. Ελπίζουμε ότι το καθεστώς ενιαίων ενισχύσεων θα διατηρηθεί. Το ερώτημα είναι γιατί πρέπει να παραιτηθούμε από κάτι το οποίο λειτουργεί καλά και έτσι δείχνει ότι λειτουργεί καλά. Ιδιαίτερα όταν είναι μια σαφής και κατανοητή λύση για τους αγρότες. Εμείς πιστεύουμε ότι έτσι όπως έχει αυτό το σύστημα ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους της ίδιας της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής και ευθυγραμμίζεται απόλυτα και με τις συστάσεις του ΠΟΕ. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να θέσουμε ένα διαφορετικό ερώτημα στους αυτούς μας. Γιατί να μην επεκτείνουμε περισσότερο την ιδέα που απορρέει από το καθεστώς αυτό. Γιατί πολύ συχνά όταν μιλάμε για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, μιλάμε για απλοποίηση, αλλά στη πράξη, αν το δείτε δηλαδή από πλευρά των νέων δημοσιονομικών προοπτικών, εγώ προσωπικά δεν βλέπω εδώ πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν να μας κάνουν να ελπίσουμε ότι θα πρόκειται για απλοποίηση για τους αγρότες. Μάλλον το αντίθετο θα συμβαίνει. Μάλλον οι διαδικασίες θα είναι πιο περίπλοκες για τους αγρότες. Και τέλος, τέλος, τελευταία μου πρόταση πρόεδρε, πιστεύω πως αν αποφασίσετε να ευθυγραμμίσετε τις πληρωμές στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός θα έπρεπε να είναι μένος συνολικός μας στόχος, αλλά πρέπει να απομακρυνθούμε από την λογική της ιστορικής παραγωγής. Το καλύτερο κριτήριο είναι η χρησιμοποιούμενη γη. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ τον κύριο, τον κύριο Πομάιντα και τώρα θα δώσω αμέσως το λόγο στο δεύτερο εμπειρογνώμονα πάντοτε για το θέμα των άμεσων πληρωμών και του καθεστώτος του ενιαίου καθεστώτος πληρωμών και θα μας μιλήσει ακριβώς για την εμπειρία της Ουγγαρίας. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι, Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Είμαι μέλος του Αγροτικού Επιμελητηρίου ε, και εργάζομαι και ως Γιώργος. Ε, ήθελα να σας μιλήσω όμως για την εμπειρία μας από το Αγροτικό Επιμελητήριο, Γεωργικό Επιμελητήριο, Επιμελητήριο Γεωργίας Τροφίμων και Ανάπτυξης της Υπέδρου, που ε, συστήθηκε πρόσφατα και έχει σαν ε, κύριο χαρακτηριστικό την υποχρεωτική συμμετοχή του. Έχουμε φτάσει τώρα στις 350.000 μέρη του γεωργικού μας επιμελητηρίου της Ουγγαρίας, ενώ στο παρελθόν έχουμε μέχρι 100.000 μέλη. Λοιπόν, είναι υποχρεωτικό λοιπόν όποιος εργάζεται στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων, της παραγωγής τροφίμων δηλαδή ή της ε, βιώσιμης ανάπτυξης, να καταστεί μέλλον μέλος του Γεωργικού Επιμελητηρίου, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πλέον προσλάβει στην Ουγγαρία και θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας πιο δυνατά και στο διεθνή χώρο. Στόχος μας είναι να στηρίζουμε τους γεωργούς, θέλουμε μια κοινή γεωργική πολιτική η οποία θα μας βοηθάει, που θα περιορίσει τις δραστηριότητε μας. Πράγμα εύκολο να το πει κανείς, αλλά είναι περίπλοκη η γεωργική πολιτική και πρέπει βέβαια να εξασφαλιστεί και η βιωσιμότητά της και η αποτελεσματικότητά της. Χρειάζεται μια κοινή πολιτική λοιπόν δίκαιη και απλή. Για δε τους κανόνες. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν να, υπάρχουν να υπάρχει ισότητα μεταχείριση σε όλη την Ευρώπη, λιγότερη γραφειοκρατία, γιατί έχουμε να κάνουμε τομεί πολύ ευαίσθητου που απαιτούν περισσότερη προσοχή. Έχουμε τομείς όπου δεν είναι απαραίτητο να ε, στοχεύουμε μόνο στην ανταγωνιστικότητα, αλλά πρέπει να κοιτάμε μακροπρόθεσμα προς το μέλλον. Και ιδιαίτερα θα αναφερθώ στην κτηνοτροφία, όπου έχουμε μόνο 35% της γεωργικής δραστηριότητας. Πρέπει να δοθεί λοιπόν περισσότερη προσοχή στους κτηνοτρόφους και στον γαλακτοπαραγωγικό τομέα. Και άλλα παραδείγματα που θα μπορούσα να δώσω. Για παραδείγματι, το τομέα των πουλερικών. Θα μπορούσα επίσης να αναφερθώ στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι νέοι γεωργοί γιατί στον πρώτο πυλώνα έχουν πολύ μεγάλη σημασία, είναι η γεωργία, αλλά θα πρέπει την υποστήριξη που προσφέρεται να την ε, έχουν στη θέση τους και βέβαια οι νέοι εισερχόμενοι στον κλάδο, αλλά και κάθε νέος γεωργός μέχρι, μέχρι 40 ετών. Γιατί πολλές φορές η αλλαγή στις γενναίες ε, στην Ουγγαρία τουλάχιστον ε, φέρνει κάποιον να μπαίνει στον τομέα της γεωργίας μετά την, ε, τα 40 χρόνια ηλικία. και άρα δεν μπορεί να απολαύσει αυτές τις ενισχύσεις που προβλέπατε για τους νέους γεωργούς για τις εκτάσεις οικολογικής καλλιεργίας. Συμφωνούμε με την αρχή. Είναι μια καλή αρχή όπως την αντιλαμβανόμαστε, την υποστηρίζουμε. Βλέπουμε ωστόσο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα διότι προτείνεται η αγρανάπευση υποχρεωτικά σε αρρώσιμες γης πολύ καλής ποιότητας. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Ε, ε, με τις τιμές που παρουσιάζονται στην αγορά και με την πείνα που επικρατεί στον κόσμο, ε, είμαστε υποχρεωμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε καλή ποιότητα αρρώσιμη γη. Με την αγρανάπευση όμως περιορίζεται πολύ σημαντικά ο αριθμός των εκτάσεων προς καλλιέργεια. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση και, προς, έκκληση και προς το Συμβούλιο και προς το Κοινοβούλιο. γιατί χρειάζονται πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για την μετάβαση. Στις επιδοτήσεις ε, της περιφερειακής ανάπτυξης. Για τις χώρες ε, οι οποίες έχουν το σύστημα και καθώς σε μια ε, θα πρέπει να πω ότι χρειάζεται να ισχύουν τα ίδια μέτρα και σταθμά για τους πάντες. Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικούς κανόνες για τους μεν και διαφορετικούς για τους δε. Θέλουμε πιο απλούς κανόνες και νομικά ε, επίσης, αλλά πάνω απ' όλα πιο κατανοητούς και ε, εύκολους στην εφαρμογή τους. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν προσεγγίζουν ε, την δυνατότητα για την ενίσχυση, γιατί είναι περίπλοκες οι διατάξεις, είναι δύσκολο να καταλάβουν τι ευκαιρίες τους ανοίγονται και είναι πολύ μεγάλο το γραφειοκρατικό άχθος. Ε, βεβαίως και πρέπει να γίνεται έλεγχος αυστηρός στα κονδύλια τα οποία διατίθενται, αλλά δεν είναι δυνατό να ξεκινούμε κακοπροαίρετα και με καχυποψία, θεωρώντας ότι ο καθένας είναι ε, ε, υποψήφιος απαταιώνας ότι προσπαθεί να σφετηριστεί ευρωπαϊκά χρήματα. Πρέπει να έχουμε μια καλοφέρετη προσέγγιση. Όλα αυτά λοιπόν είναι προσεγγίσεις, προσεγγίσεις κοινέ σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό και θα πρέπει τα προβλήματά μας, ε, ό,τι προβλήματα υπάρχουν, να έχουμε ευκαιρία να δούμε εδώ. Γι' αυτό και σας τα ε, εξέθεσα τα προβλήματα που έχουμε ε, εντοπίσει εμείς. Αν υπάρχουν ε, σημαντικές ε, ερωτήσεις, πολύ ευχαριστώ να απαντήσω. Στο βαθμό που μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ γιατί τηρήσατε το χρόνο που σας έδωσα. Λοιπόν, ξεκινάμε συζήτηση για αυτές τις δύο παρεμβάσεις. Έχει ζητήσει το λόγο ο Αντιπρόεδρος Κυριέσκη. Εάν θέλει κάποιος άλλος το λόγο να μου το πει. Παρακαλώ. Δεν ήθελα να είμαι ο πρώτος που θα πάρει το λόγο, αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Ένα γενικό σχόλιο. Μιλάμε εδώ για τις εμπειρίες των νέων κρατών μελών που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πιστεύω και νομίζω πως αξίζει να αναλυθούν εις βάθος. γιατί έτσι θα μπορούσε να ε, εμπλουτιστεί η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ακούσαμε δύο παρουσιάσεις μέχρι στιγμής, τις βρήκα και τις δύο πολύ ενδιαφέρουσες και νομίζω πως θα μπορούσαμε να πούμε ότι πάντοτε ε, είναι φυσικό να έχει κανείς εθνική προσέγγιση ακόμα και όταν είναι επιστήμονας επηρεάζεται. Και γι' αυτό πιστεύω πως θα ήταν ε, σκόπιμο να καλέσουμε εμπειρογνώμονες και εκτός, ώστε να δουν με πιο αντικειμενικά τις αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτά τα κρατη Είναι κρίμα που δεν ακούσαμε μια τέτοιου τύπου ανάλυση. Έγιναν διάφορες αναλύσεις στην προεταξιακή φάση. Αλλά νομίζω πως το ενδιαφέρον κάπως έχει ε, μειωθεί. Όταν μιλάμε για διαέβρεση, κατά κάποιο τρόπο είμαστε κάπως μπλαζέ σε σχέση με αυτό το θέμα. Έγινε η διεύρυνση και έγινε σε μια φάση όπου υπήρχαν κάποια χρήματα για την Γεωργία, πράγμα το οποίο μάλλον υπήρχαν χρήματα ε, λιγότερα από ότι τελικά είχαν υπολογιστεί αρχικά από τις αναλύσεις που έγιναν στην προενταξιακή περίοδο. Αλλά φυσικά ε, λειτουργούν διάφορες δυνάμεις της αγοράς εδώ. Έχουμε αλλαγές, για παράδειγμα, στους δασμούς, στα τέλη, στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Και όταν η Πολωνία προσχώρησε στην Ένωση, ήταν εντελώς νέα στην αγορά. Ήταν τελείως νέα η κατάσταση. Φυσικά και προσπαθούσαμε να ανοίξουμε και παλιότερα ε, τις αγορές μας, αλλά υπήρχαν πολλοί φόβοι από πολλές ομάδες της κοινωνίας μας και οι επιπτώσεις ήταν ε, τεράστιες και για τον Πολωνό αγρότη. Όλα αυτά πιστεύω πως εξακολουθούν να ισχύουν. Επίσης, ε, νομίζω πως πρέπει να κατανοήσουμε πως οι οικονομίες των νέων κρατών μελών είχαν πολλά να κάνουν για να περάσουν από τις ε, κεντρικά ελεγχόμενες οικονομίες στην ελεύθερη αγορά. Διότι παλιότερα η Γεωργία ελεγχόταν και αυτή από την κεντρική από τον κεντρικό έλεγχο και η γεωργία ήταν ε, κοινωνικό και εκτιμένο σε βαθμό 80%. Είχαμε μόνο κάποιες, ε, εκείνες τα τεράστια εθνικά ε, αγροκτήματα, είχαμε συνεταιρισμούς, αλλά η συμμετοχή στους συνεταιρισμούς ήταν υποχρεωτική. Στην ουσία αναγκαζόσουν θελοντικά να συμμετέχεις. Όπω καταλαβαίνετε τα πράγματα άλλαξαν ε, δραστικά. Ο κόσμος ωστόσο έχει στο μυαλό του εκείνες τις εμπειρίες, ε, ότι αναγκάστηκαν δηλαδή να συνεργαστούν και να συμμετέχουν σε κάτι γιατί αυτό ήταν το μοντέλο που τους είχε επιβληθεί. Και ξέρω πως ε, εμείς και πολλά άλλα κρατημέλη έχουν αυτό στο μυαλό. Είχαμε εκείνα τα κουπόνια με τα οποία αγοράζαμε τρόφιμα. Δεν υπήρχαν αρκετά τρόφιμα στην Πολωνία. Ε, χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια λοιπόν για να αλλάξουμε αυτό το σύστημα, αλλά αποφασιστικότητά μα ήταν τέτοια που πιστεύω ότι πολλοί δεν την καταλαβαίνουν, δηλαδή πολλοί κόσμοι εκτός των χωρών αυτών. Και η αποφασιστικότητα αυτή δεν αντιστοιχεί στην αποφασιστικότητα των κρατών που τώρα θέλουν να μπουν στην Ένωση γιατί το σημείο εκκίνησης μας ήταν ένα ε, σημείο απόλυτης στόχιας. Δεν είχαμε άλλη επιλογή, αν θέλαμε δηλαδή να βγούμε από αυτή τη φρικτική κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ συγκεκριμένο το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργήσαμε. Και εγώ ήμουν υπεύθυνος για τα θέματα ε, της τρεματικής ενίσχυσης στο Υπουργείο της Πολωνίας και εμείς επιλέξαμε τις πληρωμές ένα εκτάριο τότε. Ξέραμε ποιες ήταν ε, οι επιπτώσεις. Ξέραμε τι συνέβαινε στον ΠΟΕ και αυτό το ανέφερε ο κύριος Πομάιντα. Δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε δηλαδή στο δρόμο των συνδεδεμένων πληρωμών, όπου δηλαδή οι πληρωμές εξαρτώνται από την παραγωγή. Ε, τα μεγάλα αγροκτήματα ίσως να ζημιώθηκαν λόγω της αποφασής μας, αλλά τα κοινωνικά αγροκτήματα βοηθήθηκαν έτσι. Θα μπορούσε δηλαδή κανείς να πει πως ε, η προσέγγιση αυτή λειτουργήσε. Ναι, ναι, θα ολοκληρώσω. Όσο μιλάμε περισσότερο για την μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, τόσο περισσότερο αμφιβάλλω για το κατά πόσο θα πρέπει να διατηρηθεί μόνο η στρεματική πληρωμή. Εγώ πιστεύω πως αυτός ο τρόπος θα πρέπει να είναι μόνο ένας από τους τρόπους ενίσχυσης προς τους γεωργούς. Όμως η Γεωργία διαφέρει σε ολόκληρη την Ένωση ε, και πρόσφατα διαφοροποιήθηκε ακόμη περισσότερο μετά από τη διεύρυνση και θα πρέπει πιστεύω να λάβουμε υπόψη αυτήν ε, την ποικιλομορφία της Γεωργίας. Και εν γέννη να πω ότι η κοινή γεωργική πολιτική λειτουργεί αρκετά καλά κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ. Κύριε Δες, ευχαριστώ πολύ. Με χαρά παρακολουθώ τις εξελίξεις στα νεα κρατημέλη κράτη-μέλη και εγώ τα επισκέπτομαι συχνά είτε είναι Πολωνία, είτε είναι Ουγγαρία, Λετωνία, Λετωνία και με, πολύ, με εντυπωσιάζουν πολύ ε, οι επιδόσεις και οι προσπάθειες των γεωργών στις περιοχές αυτές. Είτε είναι μεγάλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, είτε μικρές, βλέπω πόσο μεγάλη είναι η προσφορά των, των οικογενειών που εργάζονται. Και, και οι δύο λοιπόν εμπειρογνώμονες μας είπαν ότι ε, θα ήθελαν απλούστευση των ε, διαδικασιών. Αλλά νομίζω ότι δυστυχώς οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν διευκολύνουν προς το στόχο αυτόν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε στη συνεργασία με το Συμβούλιο να εξυπηρετήσουμε και να ε, υλοποιήσουμε το στόχο. Αλλά πρέπει να συνεργαστούν και τα κράτη-μέλη. Χθες το βράδυ κοίταξα μαζί με τον, με τον ε, γιο μου ε, τις αιτήσει που έχουν κατατεθεί ε, φέτος, ε, που είναι η πρώτη χρονιά όπου δεν έχουμε ιστορική αναφορά. Δεν υπάρχουν πλέον στη Γερμανία συνδεδεμένες ενισχύσεις ε, και, και βέβαια αυτό οδηγεί σε μεγάλη απλούστευση. Απλώς καταγράφεται η έκταση, τα εκτάρια δηλαδή, ή καλλιέργεια, το είδος της καλλιέργειας και έτσι ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα η υποβολή της αίτησης για την ε, ενίσχυση. Λυπούμε όμως ε, για το ότι δεν έχουμε μπορέσει να προχωρήσουμε σε μια εξίσωση ανά την Ευρώπη αυτών των ενισχύσεων πιο γρήγορα. Γιατί αν δούμε τι είδους ποσά καταβάλλονται σε ενισχύσεις ανά εκτάριο και κυρίως για τα περισσότερα από τα νέα κράτη-μέλη είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε να κάνουμε με αδικία. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκα και την ε, Ουκρανία ως ε, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, αντιπροσωπείας και βλέπω ότι και για την Πολωνία και τα λοιπά καινούρια κράτη της Ευρώπης και για την Ουκρανία υπάρχουν πολύ μεγάλες βέβαια εκμεταλλεύσεις, αλλά και πολλές οικογενειακής ε, οργάνωσης εκμεταλλεύσεις. οι οποίες χρειάζονται ενίσχυση. Και από ό,τι μαθαίνω δεν έχουν καμία κρατική επιδότηση οι Ουκρανοί γεωργοί, ακόμα και οι πιο μικρές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ε, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα προβλήματα και στην Ουκρανία είναι πολύ μεγάλα, πολύ μεγαλύτερα από ό,τι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Ο κύριος Σικέρσκι αναφέρθηκε στην ε, σχεδιασμένη οικονομία. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτά. Πολλές φορές στην ε, ιδιαίτερη μου πατρίδα, όπου έχω να συζητήσω διάφορα ζητήματα επιλογών της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής των ευρωπαϊκών οργάνων, βρίσκομαι αντιμέτωπος με το δίλημα σχεδιασμένη οικονομία ή όχι. Και μάλιστα τις προάλλες στον Κουρέα, ε, είχα μια συζήτηση όπου μου έλεγε ότι ε, υπάρχουν προδιαγραφές για το πόσο μακριά θα πρέπει να είναι η τρίχα που κόβεται ώστε όταν πέφτει κάτω και συλλέγεται με το σάρωτρο να μην είναι υπερβολικά μεγάλη και ενοχλεί τον ε, πελάτη. Ε, τέλος πάντων, αυτά όλα με οδηγούν σε σκέψεις για τη σχεδιασμένη οικονομία που λέγαμε, ε, για πράγματα τα οποία δεν εξυπηρετούν βέβαια το στόχο της απλούστευσης. Ευχαριστώ κύριε Μαγκίνες τώρα. Ευχαριστώ. Και συμφωνώ με τα σχόλια του κύριου και εγώ. Με ενδιαφέρον άκουσα δύο μηνύματα που μας ήρθαν από τους προσκεκλημένους μας, που λένε ότι θέλουν να διατηρηθεί το σύστημα της ενιαίας τραματικής ενίσχυσης στην μεταρρύθμιση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας στις διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα όμως να ακούσω περισσότερο όσον αφορά τις επιπτώσεις από τις πληρωμές της κοινή γεωργικής πολιτικής στις δύο χώρες. Δηλαδή, τι επιπτώσεις έχουν οι πληρωμές αυτές στην παραγωγή. Αυξήθηκε, μειώθηκε, οι εισοδιέ αυξήθηκαν ή μειώθηκαν. Τι έγινε στην Ήπεθρο, τι έγινε με την δομή των ε, μονάδων. Γιατί πρέπει να δούμε περισσότερο με λεπτομέρειες και να ξέρουμε σε επίπεδο ακριβώς ε, αγροτικών εκμεταλλεύσεων τι αλλάζει. Αν έχετε τέτοιες πληροφορίες θα ήταν πολύ σημαντικό να μας τις δώσετε. Επίσης, οι δύο ειδικοί εδώ θα ήθελαν να μου πούνε αν έπρεπε να απομακρυνθούν από το σύστημα ενιαίας ενίσχυσης το κόστος μας είπε 4,5% ε, αν αλλάζαμε εντελώ και πηγαίναμε σε ένα νέο σύστημα, πόσο θα κόστιζε αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους εισηγητές και στους δύο για μια σύντομη απάντηση στις ερωτήσεις και μετά θα περάσουμε στο επόμενο τμήμα της συζήτησης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να ευχαρίστω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας πω ότι ήταν κάπως λεπτομερής και ίσως να μην είμαι σε θέση να απαντήσω τώρα πλήρως. Αλλά ο καθηγητής Ζεύσκη, ο οποίος θα μιλήσει αργότερα, σίγουρα θα αναφερθεί σε μερικά από αυτά που ρωτήσατε. Εγώ αναφέρθηκα στο κόστος το διοικητικό που πληρώνει τώρα η Πολωνία σε σχέση με το καθεστώς ενιαίας τραυματικής ενίσχυσης, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Δεν μιλούσε για το βάρος. Το μέσο όρο του διοικητικού κόστους, που σας είπα ότι για κάθε αίτηση είναι 100 ευρώ. Αν έχετε 1,4 εκατομμύρια αιτήσει το χρόνο, το υπολογίζετε εύκολα και βλέπετε πόσο μεγάλα ποσά πληρώνουμε. Και το μεγαλύτερο μέρος έχει να κάνει με τις επιθεωρήσεις και την συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής. Δεν μπορώ να σας πω εδώ και τώρα τι αλλαγές θα είχαμε στο κόστος εάν αποφασίζαμε ένα νέο σύστημα. Γιατί θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή με το νέο σύστημα. Και σίγουρα θα έπρεπε κάπως να το δουλέψουμε για να υπάρχει πολλαπλή συμμόρφωση και με τις ε, Ευρωτικέ περιοχές που παίρνουν την ανάπτυξη κλπ. Θα χρειαζόταν δηλαδή πολύ μεγάλη ανάλυση, τεράστιοι υπολογισμοί και αν έπρεπε να το κάνει αυτό η Πολωνία θα το έκανε, αλλά θα έπρεπε να περιμένουμε πρώτα την απόφαση για να το υπολογίσουμε. Μια προετοιμασία έτσι κι θα κόστιζε πολύ. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Πάντως προς το παρόν ευτυχώς οι συζητήσεις στην Πολωνία ε, πάνε προς το ότι θα διατηρηθεί το καθεστώς ενιαίας τραυματικής ενίσχυσης. Τουλάχιστον στην Πολωνία αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Ευχαριστούμε. Ζόφι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω κι εγώ σε κάποιες ερωτήσεις και να διευκρινίσω κάτι που να ήταν σαφές από την παρέμβασή μου. Ότι δηλαδή εμεί δεν επιδιώκουμε την διαφύλαξη του και σε επαόριστον. Δεν είναι αυτό ο στόχος μας. Η Ουγγαρία δεν επιδιώκει πάση θυσία την ε, διαθετήρηση του ΚΕΣΕ. Απλώς θέλουμε να δούμε πώς θα εξασφαλιστεί η μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο και πώς θα εφαρμόζεται στο μέλλον αυτό. Πιστεύουμε ότι το πιο σημαντικό κόστος δεν θα είναι το κόστος της μετάβασης της ίδιας. Αλλά το γεγονό ότι δεν είναι σαφής οι δομές ακόμη, γιατί είναι πολύ, πολλά τα νομοθετήματα που βρίσκονται υπό επεξεργασία, υπό προετοιμασία, και δεν μπορούμε να έχουμε τι απαντήσει που χρειαζόμαστε. Για δε την παραγωγικότητα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακή κλίμακα. Πρέπει να τις υποστηρίξουμε βέβαια. Είναι προφανές αυτό. Πιστεύουμε ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αν δεν ε, λάβουν ενίσχυση, δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν, δεν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ε, βιωσιμότητά τους και μια αποδεκτή ε, παραγωγικότητα. Εάν θέλουμε όμως να παραμείνει ο κόσμος στην Ήπεθρο, θα πρέπει να στηρίξουμε τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Η Ουγγρική κυβέρνηση λοιπόν πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι κατά 50% ιδιοκτησία των μεγάλων εκμεταλλεύσεων, οι αερόσιμες γέες. Το υπόλοιπο μόνο εκεί στις μικρότερες εκμεταλλεύσεις. Ε, αυτή η δομή πρέπει να αλλάξει. Και ελπίζουμε ότι με τη νέα νομοθεσία θα συμβάλλουμε στην εξέλιξη αυτή. Και ελπίζουμε να μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτές τις, ε, αυτά τα νομοθετήματα που είναι απαραίτητα για να αλλάξει η κατάσταση με ειδική πλειοψηφία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτό την πρώτη συζήτηση και περνάμε σύντομα στην επόμενη, στο δεύτερο τμήμα που αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου. Οι συγητές μας είναι η κυρία Ελίτα Μπέγκα που είναι επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξης Υπαίθρου του Λετωνικού Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και θα μιλήσει για το πρόγραμμα στήριξης για την ανάπτυξη υπαίθρου, δικαιούχη και κατάσταση του γεωργικού τομέα. Και στη συνέχεια έχουμε την κυρία Εμίλια Μοχάν που είναι υφυπουργός Γεωργίας της Ρουμανίας αρμόδια επί των ευρωπαϊκών υποθέσεων και θα μα μιλήσει για την ενίσχυση τη υποπεριφερειακή οικονομία μέσω των νέων πολιτικών τη κοινή γεωργική πολιτική για του μικρού καλλιεργητέ Ρουμανία. Παρακαλώ, κυρία Ελίτα Μπέγκα, για 10 λεπτά. Ε, Κυρίε και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνω την παρουσίαση για την κατάσταση στην Λετωνία όπως θα ακούσετε, εκπροσωπώ το Ινστιτούτο Γεωργικής Οικονομίας της Λετωνίας, το οποίο αξιολογεί τα προγράμματα από το 2007 στο το 2013. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τώρα τα αποτελέσματα των μελετών μας αυτά τα πέντε χρόνια που εισήχθη το πρόγραμμα περιφερειακής ε, ανάπτυξης πέθρου. Είχαμε 113.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις με 708.000 ε, περίπου ε, πληθυσμό που αντιστοιχούσε αυτές τις εκμεταλλεύσεις. Είχαμε μια στόχευση τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στη γεωργία και τη δασοκομεία, γενικά της ευημερίας της ε, περιοχής Υπέθρου, με τέσσερις άξονες, την ανταγωνιστικότητα, ο πρώτος, το δεύτερο, ο δεύτερος άξονας είχε να κάνει με το περιβάλλον και τη βελτίωση της υπαίθρου. Τρίτος, βελτίωση της ποιότητας ζωής και διαφοροποίηση. Και τέταρτος, προσέγγιση του προγράμματος LEADER. Η Λετωνία είναι από τα λίγα κράτη που έχει ε, εφαρμογή του προγράμματος Λίτερ σε ολόκληρη την έκτασή της, με πολύ μεγάλη συμμετοχή και τεράστια σημασία του προγράμματος αυτού για τη Λετωνία. Μπορεί να μην ε, ε ότι έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στην γεωργική παραγωγή το πρόγραμμα Λίτερ, αλλά ιδιαίτερα για την ανάπτυξη πέθρου έχει τεράστια σημασία. Τώρα τα δεδομένα δείχνουν για το 2010 μία μείωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 83.000 με πληθυσμό 651.000. Πάλι συνήκνονται δηλαδή ο πληθυσμός στην περίοδο αυτή. Μια εξέλιξη την οποία αντίστοιχα παρατηρούμε και σε άλλες χώρες. Εμείς περιμέναμε να παραμείνουν περισσότεροι κάτοικοι στις περιοχές υπαίθρου, αλλά δεν συνέβη αυτό. Τώρα το πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης και κατανομή των κονδυλίων. Είναι πολύ σημαντικό για την ε, Λετωνία να έχουμε ε, τα κονδύλια για την ανταγωνιστικότητα 38% στην αρχή 42% περίπου μετά ε, μετά έχουμε επίσης διατήρηση των ενισχύσεων στις εκτάσεις με αύξηση των ποσών αυτών για τις περιοχές αυτές και ποσοστά για την διαφοροποίηση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Εδώ μπορείτε να δείτε την κατανομή των κονδυλίων ανά εκμετάλλευση. Στο μπλε χρώμα βλέπετε ποσοστιαία εκπροσώπηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που είναι κατά συντριπτικό ποσοστό μικρέ στη Βετονία και στο δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρί ενίσχυση. Η υποστήριξη όμω είναι πολύ μικρή για τι ε, εκμεταλλεύσεις αυτέ, είναι περίπου στο 5% του συνόλου των ενισχύσεων. Οι μεγάλε εκμεταλλεύσεις έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό των κονδυλίων, άρα ενισχύουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους σε μεγάλες ε, επιχειρήσεις και άρα μπορούν να είναι ανταγωνιστικές και σε διεθνές επίπεδο με παραγωγή σιτηρών κτλ. Ενώ οι μικρές ε, εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Εάν κοιτάξουμε την Ευρώπη στο σύνολό τη, στο βορρά και την Ανατολική Ευρώπη, στο σκούρο μπλε χρώμα, έχουμε ένα ποσοστό 5% στην χρήση της γης για σιτηρά, καλλιέργεια σιτηρών. Πρόκειται για περιοχές οι οποίες θα προμηθεύσουν ολόκληρο τον κόσμο στα επόμενα χρόνια, θα διαθέτουν τα σιτηρά τους, τα τρόφιμα γενικά, σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ βλέπετε διαφορές μεταξύ των ε, κρατών της Λετωνίας και των κάτω χωρών. Στο δεξιά βλέπετε ότι έχει πολύ καλές προοπτικές η Λετωνία ως προς τις εκπομπές διοξιδίου, ε, μάλλον αερίων του Οι κάτω χώρες βρίσκονται σε δύσκολη θέση, ενώ η Λετωνία έχει πολύ καλές επιδόσεις. Εάν δούμε τώρα αντίστοιχα μία προβολή σε παραγωγή ενός εκατομμυρίου ευρώ στο αριστερό γράφημα, η Λετωνία έχει πολύ χειρότερες επιδόσεις από ό,τι κατά χώρες. Άρα ε, το κριτήριο αυτό των εκπομπών μπορεί να το δει κανεί ε, από διαφορετική σκοπιά και να δώσει διαφορετικά αποτελέσματα. Εάν είχαμε δηλαδή ποσοστώσει αντίστοιχε με αυτέ ε, των άλλων κρατών, θα ήμασταν πολύ λιγότερο ανταγωνιστικοί. Ενώ τώρα φαινόμαστε ω ένα κράτο πολύ οικολογικό και πράσινο. Ε, αν ακολουθήσαμε τις ποσοστώσεις των άλλων κρατών, θα χάναμε σημαντικό ποσοστό ανταγωνιστικότητας. Εδώ βλέπετε λοιπόν τον άξονα της ανταγωνιστικότητας και το τι έχει προσφέρει στην γεωργία. Το 75% όλων των επενδύσεων στη γεωργία, 376 εκατομμύρια περίπου, έχουν αξιοποιηθεί στο χώρο της γεωργίας. επενδύσεις στις υποδομές, επενδύσεις στην ε, κατεργασία τροφίμων, ε, βελτίωση της οικονομικής αξίας ε, και λοιπά μέτρα που έχουν το 7% περίπου στο μπλε χρώμα. Ποσοστό απασχόλησης τώρα στη Λετωνία. Εδώ βλέπουμε λοιπόν κάποιες ε, εξελίξεις σε σχέση με τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αξίες παραγωγής, αν ε, λάβουμε ως κριτήριο δηλαδή την αξία της παραγωγής, έχουμε ένα 9,3% των εργαζομένων που θα χρειαστούν για την εξασφάλιση του ίδιου ε, παραγόμενου προϊόντος άρα χρειάζεται βελτίωση ανταγωνιστικότητα. Εδώ έχουμε ένα γράφημα το οποίο πόσο, δείχνει πόσο καλά έχουμε αντιμετωπίσει την κρίση. Με σημαντική αύξηση των τιμών των γεωργικών προϊόντων, όπως και των εσόδων, μπορεί να έχει μειωθεί ελαφρά ο αριθμός των ε, εργαζομένων, αλλά η παραγωγικότητα δεν έχει πληγεί και ε, δεν έχει πληγεί το γεωργικό εισόδημα. Οι μακροβρόθεσμες επενδύσεις είναι μικρότερες. Οι προοπτικές Το εσόδων είναι σε επίπεδο καλό όμως, γιατί μειώθηκαν οι επενδύσεις μέχρι το 2010 και μετά παρουσιάζουν άνοδο. Το γεωρικό σύνδεμα παρουσιάζει άνοδο. έχουμε περίπου 6.000 ευρώ εισόδημα ανά στη Γεωργία. Ποσοστό από τα χαμηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δείχνει ότι έχει περιθώριο για βελτίωση ακόμη περισσότερο της ανταγωνιστικότητάς της η Λετωνία. Σε αυτό θέλω να πω ότι είναι πολύ διαφορετικές οι καταστάσεις που παρουσιάζουν τα κράτη-μέλη ανάλογα με τη στάση του καθενό, η, η ε, κατάσταση του περιβάλλοντος, παραδείγματι, στην ε, γεωργία και την, ε, τις κάτω είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με αυτό που σημειώνεται στην Λετωνία. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση και παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας της Ρουμανίας, την κυρία Εμίλια Μοχάνου να λάβει το λόγο. Έχει το λόγο, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσω σύντομα να σας εξηγήσω πώς η μικρή Γεωργή στη Ρουμανία γιατί βέβαια και υπάρχουν μικροί γεωργοί, πώς εισπράττουν λοιπόν αυτές τις ενισχύσεις χάρη στις πολιτικές που έχει εισαγάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα θα συγκρίνω λίγο δύο περιόδους. 1989 και 2012. Τι είναι το σημαντικό τώρα στη σύγκριση αυτή. Το βλέπετε στη διαφάνεια. 13,7% εκτάσεις. Ήταν κατανεμημένες σε ένα 28% των γεωργών που είχαν εντατική ε, παραγωγή και οι υπόλοιποι είχαν ε, εκτατική. Όπου είχαμε 3.386 ε, τέτοια καθεστώτα ενιαίας τραυματικής ενίσχυσης. Τα 14,7 εκατομμύρια όμως περιορίστηκαν σε 9,7. 12.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις με εντατική καλλιέργεια και 900.000 εκτατικής. 3 εκατομμύρια εκτάρια. Υπήρχαν βέβαια και κάποιες και υπάρχουν μεσαίες εκμεταλλεύσεις που καλύπτουν 1,7 εκατομμύρια εκτάρια. Και υπάρχουν ακόμα 2 εκατομμύρια εκτάρια τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο καθεστώς ενιαίας τραυματικής ενίσχυσης. Εδώ νομίζω ότι βλέπετε καλύτερα το ότι υπάρχει μία συγκέντρωση των ε, εκμεταλλεύσεων, των πιο μικρών, αν τη συγκρίνουμε με τις πιο μεγάλες, οι οποίες μερικές φορές είναι και 16.000 εκτάρια. Εδώ τώρα τι μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει το πρώτο τμήμα του γραφήματος αυτού, όπου βλέπουμε ότι οι μικρές ε, εκμεταλλεύσεις, 1 έως 10 εκτάρια, είναι πάνω από 90% των συνολικών εκμεταλλεύσεων. Και στην πραγματικότητα εκμεταλλεύονται μόνο 15% της επιφάνειας που περιλαμβάνεται στο ΚΕΣΕΠ. Αν τώρα ε, δούμε πιο συγκεκριμένα τις ε, εκμεταλλεύσεις ενός 10 εκτάρια, εδώ βλέπετε από τα στατιστικά ε, δεδομένα που έχουμε, ότι πρόκειται για έναν μεσαίο αγροτικό χώρο όπου διαπιστώνονται θετικά και αρνητικά στοιχεία. Υπάρχουν δύο περιφέρειες, το κόκκινο και στο ροζ, όπου έχουμε πολύ λίγες μικρές εκμεταλλεύσεις. Και αυτό συμβαίνει γιατί πρώτα απ' όλα εκεί βρίσκεται το Βουκουρέστι, πρωτεύουσα. Οπότε εννοείται εκεί πρόκειται για μια αστική περιοχή, μια πόλη, όπου έχουμε φυσικά τον ε, μικρότερο αριθμό ε, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η άλλη περιφέρεια βρίσκεται στα σύνορα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν είναι ανταγωνιστικός ο αγροτικός τομέας σε θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι μερικές φορές κάποιοι αγρότες καταλαμβάνουν έναν χώρο που κανονικά θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος πολύ πιο αποδοτικά. Πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι η βιοπικιλότητα και το περιβάλλον είναι πράγματα τα οποία παραδοσιακά λαμβάνουμε υπόψη μας στη Ρουμανία, όπως επίσης το θέμα του τοπίου, της προστασίας του τοπίου, ο αγροτουρισμός. Είναι και αυτά στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να διατηρήσουμε την γεωργία στην περιοχή, για να μην μάλιστα μερικές φορές μπορούν έτσι και να επιτρέψουν οι αγρότες τη γη τους. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω τις λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ε, με τον κομμουνισμό καταστράφηκαν πάρα πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και πολλοί συνεταιρισμοί. Υπονομεύθηκε τότε κάθε προσπάθεια ιδιωτική πρωτοβουλίας, κάτι το οποίο ευτυχώ δεν είναι έτσι σήμερα οι πιο μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημογραφία, διότι επιτρέπουν να αποφύγουμε την απομάκρυνση του πληθυσμού από την περιφέρεια. Τώρα πόσο βιώσιμες είναι οι εκμεταλλεύσει αυτές. Από τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε, ξέρουμε ότι ο κύριος πόρος για τις οικογένειες που απασχολούνται εκεί είναι η γεωργία, 37,6% δηλαδή του συνόλου των εσόδων τους. Το μεγαλύτερο ε, μέρος βέβαια έχει να κάνει με την κατανάλωση των ε, δικών τους προϊόντων. Και μόνο 9% είναι αυτό που ξοδεύουν σε χρήματα. Τι συμπέρασμα πρέπει να βγάλουμε από όλα αυτά ότι δεν είναι πρόβλημα αυτές οι μικρές εκμεταλλεύσεις στη Ρουμανία. Τα έσοδα είναι πολύ χαμηλά, όπως έλεγε και ο προλαλής σας. Ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της παραγωγής είναι κάτι πάρα πολύ περιορισμένο σε αυτές τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Από την άλλη βέβαια το γεγονός ότι στην Ήπεθρο, στη Ρουμανία έχουμε πολύ χαμηλότερη ανεργία από ότι στις αστικές περιοχές αποτελεί ένα δίκτυο ασφάλειας για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης και για νέες επίσης, για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Κάτι άλλο το οποίο βλέπουμε είναι οι ηλικιωμένοι σημαντικό ποσοστό ε, των ανθρώπων που ζουν στις αγροτικές περιοχές είναι πάνω από 50 ετών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε νέους αγρότες να μπουν στην γεωργική δραστηριότητα. Και πρέπει επίσης να προβλέψουμε και να σκεφτούμε ότι η αύξηση στην ανταγωνιστικότητα δεν πάει σε συνάρτηση με το μέγεθος μιας γεωργικής εκμετάλλευσης καθόλου. Έχουμε πολλά παραδοσιακά προϊόντα. Έρχομαι τώρα στην αναδιάρθρωση. Η οικονομική διάσταση με εμπορική διάσταση είναι κάτι που πρέπει να ενισχύσουμε πρέπει να στηρίξουμε την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και να εκπονήσουμε πολιτικές οι οποίες επιτρέπουν στους αγρότες να επιλέξουν το μέλλον τους. Να τους στηρίξουμε χωρίς να μπλοκάρουμε τον φυσικό τρόπο εξέλιξής τους. Είχαμε 900.000, είπαμε, εκμεταλλεύσεις οι 50.000 έχουν κάποιο συγκεκριμένο προσανατολισμό. Μέσος όρος 4-5 εκτάρια. Αυτό σημαίνει επίσης ότι Μάλλον πρέπει να ξέρετε επίσης ότι πολλές από αυτές οι εκμεταλλεύσεις έχουν ε, και ζώα μέσα, έχουν δηλαδή και εκτινοτροφικέ δραστηριότητες. Θα έρθω τώρα σε κάποια μέτρα τα οποία προβλέπουμε και πώς πιστεύουμε ότι τα μέτρα αυτά θα μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε με τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Για τον πρώτο πυλώνα, η άμεση στραματική ενίσχυση. Μετά για το θέμα της ζωικής ε, εκμετάλλευσης, εκεί έχουμε χαμηλά ποσοστά. Θέλουμε να ενισχύσουμε την εγκατάσταση νέων γεωργών, νέων σε ηλικία, να στηρίξουμε ομάδες γεωργών, την ε, κατάρτισή τους και να στηρίξουμε και τις μειονεκτικές περιοχές, απομακρυσμένες, βουνά κλπ. Ποιες είναι οι τάσεις τώρα που έχουμε διαπιστώσει. Πρώτον, οι διάφορες πολιτικές, προεδρυξιακές και στη συνέχεια, έχουν σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ένα-δύο εκτάρια και να αυξηθεί το μερίδιο των μεγαλύτερων τρία-τέσσερα εκτάρια να εκμετάλλευση. Με μέτρα στήριξης της υπαίθρου πάντως μπορούμε να πούμε είναι το μέτρο 141 στήριξη των μεσαίων εκμεταλλεύσεων όπου είχαμε μεγάλη ζήτηση. Οι ακρότες αρχίζουν να επικεντρώνονται στην αγορά και να διαφοροποιούν την παραγωγή τους. Θα μπορούσα να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά το μόνο που θέλω να κάνω τώρα είναι να σας δείξω κάποιες εικόνες από την δικιά μου την περιοχή που δείχνουν ότι όσο μεγάλη και αν είναι η προσπάθεια που γίνεται, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε τους αγρότες στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και τις φωτογραφίες Μια εικόνα αξίζει χίλια λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς το λόγο τώρα για τη συζήτηση. Μπρατέλα. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Όταν επισκεφθήν την ε, Ρουμανία και συνάντησα Γεωργό, μου είπαν ότι θέλει η κυβέρνηση να επιβάλλει ένα νέο φόρο. Ειδικό τέλος, ειδικό φόρο που θα επιβάρυνε τον Γεωργό ε, φόρο επί του γεωργικού εισοδήματο. Και φαίνεται ότι δεν είναι η πρόθεση της ρουμανικής κυβέρνησης. να φορολογήσει τις άμεσες ενισχύσεις. Όποιος δε δεν συμμετέχει στην καταβολή του φόρου, δεν καταβάλει τον φόρο του, θα λαμβάνει λιγότερες ενισχύσεις στο μέλλον. Θα εκπίπτει δηλαδή από το ποσό της ενίσχυσης το αντίστοιχο του φόρου που δεν κατεβλήθη. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό είναι καλό σύστημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Έχουμε κάνει πολλά για να βελτιώσουμε τα επίπεδα των άμεσων ενισχύσεων στη Ρουμανία και στις χώρες της Βαλκανικής, αφού πολλοί γεωργοί βρίσκονται σε ε, δύσκολη κατάσταση. Εδώ έχουμε να κάνουμε σημαντικά ποσά για το Γιώργο. Και αν Χρειάζεται περισσότερη, περισσότερα χρήματα. Θα εισπράττει λιγότερα κάποιος άλλος γεωργός σε κάποιο άλλο κρατός μέλος. Έγιναν λοιπόν οι αλλαγές, αλλά οι αλλαγές αυτές δεν έχουν γίνει προκειμένου να επιβαρύνει με φορολογία η ρουμανική κυβέρνηση. Δεν θα γίνει δηλαδή η, κρατική, η ανίσχυστη γεωργία φορολογικά έσοδα για την ε, ρουμανική κυβέρνηση. Δεν είναι θεμητό αυτό το οποίο ζητούν και θα πρέπει αυτός ο φόρος για τις ε, κρατικές ενισχύσεις επί των, κρατικών, των γεωργικών ενισχύσεων να καταργηθεί. Είναι απολύτως αντίθετος με, τον την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ. <clears throat> Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Έχουμε κάποιον άλλον. Κύριο Πρόεδρε, έχω κάποιες ερωτήσεις. Και για την ε, υποστήριξη των γεωργών. αλλά και για αυτό που είπατε για την υποστήριξη των ε, προγραμμάτων από προγράμματα για τους ε, νέους γεωργούς τι είδου ε, μέγεθο γεωργική εκμετάλλευση θα συνιστούσατε σε ένα νέο γεωργό ή συνιστάτε σε ένα νέο γεωργό που θέλει να ξεκινήσει μια γεωργική εκμετάλλευση, τι θα ήταν το καταλληλότερο μέγεθο επιχείρηση ε, γεωργική. Και δεύτερον, που μάλλον θα ε, έπρεπε να το χωρωτήσει το πρώτο κομμάτι των παρεμβάσεων, υπάρχουν περιοχέ στα νέα κράτη-μέλη, οι οποίε είτε δεν εντάχουν στο ΚΕΣ, είτε δεν είναι καταγεγραμμένες ε, με κάποιο τρόπο. Όπως οι παραδείγματι μισθωμένες για στη Ρουμανία που είναι αρκετά αρκετές εκτάρια από ό,τι ξέρουμε. Τι θα γίνει με αυτές. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα. Έχει προταθεί κάποια λύση, περιμένατε μια λύση μέσω της Ευρώπης ή θεωρείτε ότι οι γεές που βρίσκονται σε μπορούν να εξυπηρετήσουν το στόχο της ε, προστασίας της φύσεως. Και κάτι άλλο. στο κατά πόσο θα πρέπει να διατηρηθεί μια συγχρηματοδότηση από πλευρά των κρατών μελών στο δεύτερο πυλώνα. Τι θέση λαμβάνετε σε αυτό το ερώτημα, αυτό το δίλημα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βοτζιχόφσκι, έχετε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ο πρώτος η πρώτη ομιλήτρια μας μίλησε για την πρόταση εισαγωγή ε, διδικών φόρων ε, για τους αγρότες στη Γερμανία ε, και ξέρω πως και στην Πολωνία προετοιμάζει κάτι τέτοιο κυβέρνηση και οι γεωργοί ήδη διαμαρτύρονται. Σίγουρα είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα και θα επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση των γεωργών όχι μόνο στη Ρουμανία αλλά και στην Πολωνία από ό,τι φαίνεται. Για να επανέλθω στα όσα είπε η κυρία Μοχάν, ε, είπατε πως 2 εκατομμύρια εκτάρια στην Ρουμανία είναι γη που δεν ε, καλλιεργείται. Ποια είναι η σχέση με τις άμεσες πληρωμές κατά τη γνώμη σας ε, για αυτό το φαινόμενο, γιατί από την η εντύπωσή μου είναι ότι η γη που δεν είναι ε, καλλιεργημένη και τα ποσά που δίνονται για αυτή τη γη είναι δυσανάλογα προς ε, τις άμεσες πληρωμές. Δηλαδή όσο πιο χαμηλές είναι οι πληρωμές τόσο περισσότερη είναι η γη που μένει αργητή. Εσείς βλέπετε να υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα δύο αυτά ε, και η Πολωνία και η Ρουμανία έχουν χαμηλότερα ποσοστά άμεσων πληρωμών, αλλά πιστεύετε πως αυτό συνδέεται. Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, ο κύριος Ντες. <coughs> Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. λόγο, πάνω σε αυτή τη δήλωση που ακούστηκε ότι θα υπάρξει ή μπορεί να υπάρξει φορολόγηση των ε, γεωργικών επιδοτήσεων. Πρέπει να επαληθευτεί αν επιτρέπεται κάτι από το κοινοτικό δίκαιο. Και μου φαίνεται πολύ παράδοξο χώρες ε, της Ανατολικής Ευρώπης να ε, ξαφρίζουν αυτές τις επιδοτήσεις. Εμείς είχαμε πολύ μεγάλη συζήτηση κάνει στη Γερμανία ε, πάνω στην ανάγκη να παραιτηθούμε από ένα μέρος των επιδοτήσεων που πήγαιναν στους δικούς μας γεωργούς για να ωφεληθούν τα νέα κρατημέλη. Εάν όμως τώρα, οι γεωργοί των νέων κρατομέλων, εάν όμως τώρα έρχονται ε, κυβερνήσεις όπως αυτό που ακούστηκε για τη Ρουμανία να φορολογήσουν αυτές τις επιδοτήσεις ε, τις γεωργικές, πώς είναι δυνατόν να το δεχθούμε και να κατανοήσουμε τη λογική πίσω από αυτό. Η τωρινή κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, το εισάγει αυτό ή μήπω υπάρχουν και άλλες προηγούμενες κυβερνήσεις που είχαν σχεδιάσει τη φορολόγηση αυτή. Αυτό οπωσδήποτε δεν εξυπηρετεί το στόχο της πιο δίκαιης κατανομής ε, του γεωργικού εισοδήματος ε, στην Ευρώπη. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα ήθελα εγώ να προσθέσω μία. Ποιες είναι οι τάσεις που βλέπετε να, σχηματίζεται όσον, να σχηματίζονται όσον αφορά την αλλαγή του καθεστώτος της, ε, των γεών, των αρρώσιμων γεών, γιατί ξέρω ότι σε πολλές χώρες ακόμα έχουμε μπροστά μας αυτή την κατάσταση, δηλαδή την αλλαγή του καθεστώτος των γεών. Ποια είναι η γνώμη σας. Ευχαριστώ. Θα θέλατε να πάρετε το λόγο ε, με τη σειρά που μιλήσατε. Παρακαλώ. Ναι. Э, κοιτάξτε, είναι όντω ένα πρόβλημα ε, γιατί αν ε, το προτείνει και η δική μας κυβέρνηση να, φορολογηθεί, ε, να φορολογηθούν γεωργικές επιδοτήσεις, προφανώς κανείς δεν θα χαρεί. Πρόκειται για εισοδήματα των γεωργών από την άλλη και κάθε μορφή εισοδήματο ε, μπορεί να φορολογηθεί, να αποφάσει μια κυβερνήσεως αυτό. Και δε το ερώτημα το σχετικό με, την, με το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης, έχουμε περίπου να κάνουμε με 16.000 ευρώ στις μεσαίου μεγέθους ε, εκμεταλλεύσεις, γιατί δεν εξετάζεται η έκταση της γης, τα εκτάρια δηλαδή που έχει μια εκμετάλλευση, αλλά το τι μπορεί να κάνει μια εκμετάλλευση, που βρίσκεται, τι είδους παραγωγή έχει, πώς αξιοποιείται, τι είδους δραστηριότητες παρουσιάζει. Αυτό είναι το κριτήριο και βέβαια κριτήριο είναι πάντα ποια περιφέρεια ή ποια περιοχή θέλουμε να ε, βοηθήσουμε να αναπτυχθεί. Και φυσικά δεν υπαγορεύουμε σε κανέναν τι θα κάνει, απλώς δίνουμε συμβουλές, ε, ε, προτάσεις κάνουμε. Στη χώρα μας οι περισσότερες είναι ε, κατά ποσοστό 80-90% οι μικρές επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται να απογορευτεί να υπάρχουν μικρέ επιχειρήσει. Από την άλλη, έχουμε μεγάλο πρόβλημα και γύρανση του γεωργικού πληθυσμού, στο μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεών μα. Ε, και προσπαθούμε να κερδίσουμε νέου γεωργού για τη γεωργική παραγωγή για την κτηνοτροφία, για την καλλιέργεια των σιτηρών. Ε, δουλειές που χρειάζονται σκληρή ε, προσωπική εργασία κάθε μέρα, γιατί δεν μπορεί ποτέ η αδίποτε τεχνολογία να υποκαταστήσει τον γεωργό ή τον κτηνοτρόφο. Δεν μπορεί κανείς να πει δηλαδή, α, σήμερα δεν θα ε, αρμέξουμε τις αγελάδες. Δεν υπάρχει τέτοια τεχνολογία. Επομένω, χρειάζεται να έχουμε μια νέα γενιά νέων ε, κτηνοτρόφων γεωργών και ίσως χρειάζεται τα κίνητρα που θα δώσουμε να τους επιτρέπουν να δουλεύουν χωρίς ίσως να πρέπει να περνάνε 20 ώρες 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα σε σκληρή γεωργική δουλειά. Το ερώτημα είναι βεβαίως πώς θα ε, προωθήσουμε την ανάπτυξη αυτή. Θέλουμε να οθήσουμε τις μικρότερες επιχειρήσεις προς νέους κλάδους της αγοράς προς ε, καινοτόμα προϊόντα, ε, βιολογική γεωργία, ε, διαφορετικούς τομείς καταργασίας ενδεχομένω. Τομείς δηλαδή όπου μπορεί η μικρή επιχείρηση... E, okay, so I speak English if it's okay. So... Θα μιλήσω αγγλικά, αν δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσον αφορά τους ε, φόρους, ως εμπειρογνώμονας μπορώ να πω ότι δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη με αυτή την πολιτική. Ήδη δημιουργεί πολλά προβλήματα για τους γεωργούς. Ξεκίνησε σαν ε, δοκιμαστικά από την ε, κυβέρνηση της Ρουμανίας για να δει αν μπορούσε να συλλέξει περισσότερα χρήματα για τον προπολογισμό, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι τα μεγάλα αγροκτήματα που κατά κάποιο τρόπο δεν αισθάνονται τόσο πολύ το πρόβλημα της φορολόγησης για τις άμεσες πληρωμές. Το πρόβλημα αφορά περισσότερο τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. που ήδη διαμαρτύρονται, ήδη εκφράζουν τα προβλήματά τους. Δεν τους αρέσει καθόλου να βγάλουν αυτά τα χρήματα από την τσέπη τους και θεωρούν και ότι δεν είναι και δίκαιο να τους παίρνουν ακόμη περισσότερα. Η Ρουμανία, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι μια από τις χώρες όπου υπάρχει το, όπου επικρατεί το χαμηλότερο επίπεδο άμεσων πληρωμών και είναι χαμηλό ακόμα και, ε, και εφόσον είμαστε σε μια περίοδο phasing in και έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε αυτές τις ενισχύσεις από τον Εθνικό Προϋπολογισμό. Τώρα όσον αφορά τους νέους γεωργούς δεν ε, σκεφτόμαστε την επιβολή μάλλον την επιλογή του εκταρίου αλλά θέλουμε να ασκήσουμε μια επιτυχή πολιτική ώστε να προσελκύσουμε όσο γίνεται περισσότερους νέους γεωργούς στην γεωργία και κυρίως στον πρώτο πυλώνα. Και από ό,τι καταλάβαμε από τη νέα πολιτική, αυτό είναι ο βασικός στόχος, απλοποιημένο ε, σχέδιο, ώστε να μπορούν να προσελκυθούν νέοι και μικροί γεωργοί στο σύστημα. πολύ σοβαρό πρόβλημα δε που αναφέρθηκε είναι τα 2 εκατομμύρια εκτάρια και είναι χαρακτηριστικό πρόβλημα της Ρουμανίας, δηλαδή η γη που δεν καλλιεργείται, που δεν χρησιμοποιείται. Καταρχήν αυτά τα 2 εκατομμύρια εκτάρια δεν περιλαμβάνονται στο Άγιαξ. Δηλαδή δεν πληρώνει κανείς για αυτά, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτά αυτές οι γέες, ιδιαίτερα από το 2014 όταν θα απελευθερωθεί η αγορά των γεών. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν αυτές οι γέες να συμπεριληφθούν στο σύστημα. Και όπως είπε και κάποιος από τους ομιλητές, όσο περισσότερη γη μπει μέσα στο, στο σύστημα, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι πληρωμές. Δεν μοιράζεται το ποσό σε 9,5 αλλά σε 9,5 συν 2 εκατομμύρια. Και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα. Φυσικά θα μπορούσαν να μετρήσουν αυτά τα, αυτές οι γιές, γιατί οι περισσότερες είναι παρθένες γιές. Δεν είναι ε, παραγωγικές γιές. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το πρασίνισμα. Θα μπορούσε αυτό να είναι μια λύση. ωστόσο, δεν είναι και τόσο απλό να είναι κανείς πράσινος και εκεί ε, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποιοι όροι. Και μια ερώτηση για τη συγχρηματοδότηση <laughs> για τα κράτη-μέλη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, τουλάχιστον από όσο εγώ γνωρίζω με τη συγχρηματοδότηση από την πλευρά των κρατών μελών, είναι τουλάχιστον στη Ρουμανία οι περιφερειακοί προπολογισμοί είναι εξαιρετικά μικροί και τα περισσότερα προγράμματα, ακόμα και αν ε, ε, χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια, τα υπόλοιπα είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν από τον εθνικό προπολογισμό γιατί <laughs> είναι τέτοια η κατάσταση σε τοπικό επίπεδο. Και όσον αφορά τις τάσεις, ρωτήσατε ποιες είναι οι νέες τάσεις. Για τη διαχείριση και την παραγωγή στη Γεωργία πιστεύω πως για μας η επιτυχία που θα μπορούσαμε να σας παρουσιάσουμε είναι η βιολογική γεωργία που αυξάνεται. Όλο ένα και περισσότερες εκμεταλλεύσεις αλλάζουν από την συμβατική γεωργία στην οικολογική ή βιολογική γεωργία. Και αυτή είναι μια τάση για την οποία θα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Είναι δύσκολο, γίνεται σε μικρή κλίμακα ακόμη, ωστόσο τίνουμε να γίνουμε ε, χώρα εξαγωγής ε, προς την ε, Γερμανία τον Οκτώβριο ήμουν σε μία από τις πιο σημαντικές ε, εκθέσεις ε, τροφίμων και η Ρωμανία συμμετείχε και πραγματικά καταφέραμε να υπογράψουμε ένα σωρό συμβόλαια για πόλεις παραγωγής και πιστεύω πως αυτή είναι καλή η τάση. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ευχαριστώ. Κύριε για, βλέπω πως έχετε ε, άλλη μια ερώτηση. Παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, μια συμπληρωματική ερώτηση, καλύτερα μια παρατήρηση για τα πρακτικά. Στα πει, είπε ο κύριος Ντες, ε, και θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερως, γιατί είναι κάπως συγκεκριμένη η κατάσταση. Ε, βεβαίως και μπορεί ένα κράτος μέλος να επιβάλλει φόρο επί του εισοδήματος, αλλά δεν είναι συμβατό με την ε, κοινοτική νομοθεσία να φορολογούνται οι άμεσε ενισχύσει. Παρακαλώ και τη γραμματεία τη Επιτροπή μα να απευθύνει σχετικό ερώτημα στα κράτη για το τι ισχύει. Έχουμε αρκετές ε, αρμοδιότητες ε, ως προς την γεωργική, με την γεωργική πολιτική ώστε να μπορούμε να έχουμε απευθείας επικοινωνία και πάντως είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο ε, να συμβατεί με το κοινωνικό δίκαιο η φορολόγηση του γεωργικού εισοδήματος οι άμεσες ενισχύσεις ιδιαίτερα δεν είναι δυνατόν αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να ρωτήσουμε είτε τα κράτη-μέλη, αν κάποιο θέλει να δώσει πληροφορίες, είτε και την Επιτροπή των Επίτροπων να μα ενημερώσει. E, Δεν ξέρω τώρα. κατάλαβα τώρα αν αυτό ήταν ε, ερώτηση ή έκφραση άποψη. Θέλει κάποιο από του ομιλητέ μα να το σχολιάσει. Αν ναι, εγώ να προσθέσω άλλο ακόμα ένα σχόλιο ή ερώτηση από το πρόεδρο. Μιλούσατε για παραδοσιακή παραγωγή τροφίμων. Εσείς απομακρύνεστε από αυτήν την τάση. Ε, ποια είναι η αλλαγή για την οποία μιλήσατε. Γιατί μιλήσατε για μετακίνηση από τη συμβατική γεωργία στη βιολογική γεωργία. Uh, no, actually, the tradition... Όχι η παραδοσιακός τρόπος παραγωγής ξεκολουθεί να υπάρχει και έχουμε πολλές παραδοσιακές ε, εκμεταλλεύσεις που παράγουν ε, λάδι ας πούμε με παραδοσιακό τρόπο αλλά δεν είναι βιολογικές καλλιέργειες. Ε, η παράδοση λοιπόν παραμένει αλλά αναπτύσσεται και η βιολογική γεωργία. αναπτύσσονται παράλληλα, όχι σε ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μάρτιν, πολύ ήσυχο σε βλέπω. Σπάνια είσαι τόσο ήσυχο σε τέτοιου είδου συζητήσει που έχουμε. Περνάμε τώρα στο τρίτο μέρος, το κοινωνικό και οικονομικό σκέλος της συζήτησής μας. πιστεύω ότι λίγο πολύ έτσι θα καταλήξουμε και σε συμπεράσματα και σε σχέση με τα δύο άλλα θέματα που εξετάσαμε. Πρώτος μιλητής μας εδώ είναι ο κύριος Τσισεύσκη από το Πανεπιστήμιο του Πότσναν και θα μας μιλήσει για τις προσαρμογές της κοινή γεωργικής πολιτικής για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κόσμου και των αγροτών και αυτό βάσει βέβαια τις εμπειρίες που έχουμε από την Πολωνία. Εγώ δεν ξέρω, αυτή η προσαρμογή μπορεί να υπάρξει. Πράγματι, είμαστε όλο αυτιά. Σας ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένη. Είναι μεγάλη μου χαρά και σας ευχαριστώ να είμαι σήμερα εδώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μάλιστα είναι η δεύτερη φορά που έχω αυτή τη χαρά, διότι και παλιότερα είχα προσκληθεί ε, για να μιλήσω στην Επιτροπή σας για αυτά τα θέματα. που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, τώρα, λόγω χρονικού περιορισμού θα αφήσω τα αποκλειστικά πολωνικά ζητήματα κατά μέρο. Ε, μπορούμε ίσως να τα συζητήσουμε αργότερα. Πάντως κάποιοι προηγούμενοι μιλητές ε, τα ανέφεραν. Εγώ ωστόσο θα ήθελα να εστιάσω αλλού την προσοχή. Εγώ αντιπροσωπεύω εδώ την Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου του Πόσνανα. Ε, αυτό είναι λοιπόν το τμήμα το οποίο συνδέει την οικονομία με την παραγωγή τροφίμων και την κατανόηση της ε, παραγωγής τροφίμων στην μικροκλίμακα. Ως αποτέλεσμα, το, η, δική μου εισήγηση εξετάζει την κοινή γεωργική πολιτική ως σύστημα. Και Δεδομένης της εμπειρίας που έχουμε από το 2004, μπορούμε ήδη να σας μιλήσουμε για μια ανεκτίμηση που μπορεί να είναι και καθολικότερη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες του κ. Σικέρσκη, διότι εκείνος ανέφερε πως ε, οι καθολικές εισηγήσεις είναι πιο σπάνιες και ότι συνήθως επιλέγονται οι μεμονωμένες ε, παρεμβάσεις. Ε, Τώρα δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ε, αλλά πάντως όταν μιλάμε για κανονισμούς ή για μέσα, στην ουσία όταν εσείς συζητάτε τέτοια πράγματα, εσείς συμμετέχετε στον αγώνα για αλλαγή στον τρόπο σκέψης, διότι η κοινή γεωργική πολιτική, αν δει κανεί το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο μετά από το 2010, πριν το 2013, συνδεόταν ανέκαθεν με πολλές ε, συγκινήσεις, ακόμα και πολλές φορές συζητήσεις αντιφατικές ε, ε, και ε, προτάσεις λύσεων που δεν ήταν αποδεκτές από όλους. Ωστόσο μπορούμε νομίζω να τα συνοψίσουμε όλα αυτά και να βρούμε κάποιον κοινό παρονομαστή. Πρώτη πτυχή εδώ θα ήταν η σύγκρουση ανάμεσα στις ε, στην φιλελεύθερη επιλογή και στην ε, κρατική επιλογή. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι αλλαγές στα πρότυπα που είχαμε, δηλαδή τη βιομηχανική, κοινωνική βάση έχουμε προχωρήσει σε πιο κοινωνικά ισορροπημένη γεωργία. Ε, οι λύσεις που έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, ε, αν δούμε τη φιλελεύθερη επιλογή, εστιάζουν την αύξηση ε, του ανταγωνισμού πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και τέλος μετακίνηση των πόρων από τη Γεωργία σε άλλα κομμάτια δραστηριότητας η ε, μείωση των πλονασμάτων των ε, τροφίμων, η εξέβρεση των κατάλληλων ε, κονδυλίων. Από την άλλη πλευρά είχαμε την κρατική λύση, ας πούμε, που βασίζεται στον κρατικό έλεγχο η παρέμβαση και εκεί θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε ως εξή τα επιχειρήματα. Καταρχήν, η διαρροή των οικονομικών πλονασμάτων σε μη γεωργικούς τομείς. Ιδιαίτερα λόγω του γεγονότος ότι ο βασικός παράγοντας εδώ που είναι η γη θεωρείται ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί, είναι ακίνητη ακίνητος παράγοντας. Αν λοιπόν λάβει κανείς υπόψη και το σε επιπτώσεις της συνέργειας θα δείτε ότι κάποιες νέες, νέες ε, δομές μονοπωλιακού χαρακτήρα δημιουργήθηκαν στη Γεωργία. Σε κάποιες από τις συζητήσεις σας μιλήσατε επίσης για την αύξηση σε αρνητικών εξωτερικών παραγόντων Με άλλα λόγια, το κόστος δεν ε, ε, εσωτερικεύεται για να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα των οικονομολόγων. Επίσης, έχει αυξηθεί η πίεση στο κοινωνικό και στο φυσικό περιβάλλον. Και τέλος, η σύγχρονη γεωργία υποδίδει κάποια αγαθά τα οποία δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν. Αυτή είναι η σύνοψη των συζητήσεων σας μέχρι στιγμής και οι δύο αυτές οι επιλογές αντιμαχόμενες που δημιουργούν διλήμματα για τη γεωργία στην Ένωση. Επιπλέον η έννοια της νέας ε, οικονομία τη αγορά έχει δημιουργηθεί όπου οι γεωργικές βιομηχανικέ αλλαγέ, μάλλον αλλά, οι, οι, γεωργική βιομηχανία μετατρέπεται σε κοινωνικά ισορροπημένη γεωργία. Όλα αυτά επηρεάζονται και βέβαια και από άλλους παράγοντες όπως καταρχήν την ανάγκη εγγύησης κάποιων ε, κοινωνικών, ε, οικονομικών και περιβαλλοντικών πτυχών στην ε, ισόρροπα. Δεύτερον την ανάγκη αλλαγής όσον αφορά την μεταφορά οικονομικών πλεονάσματος σε μια φάση παγκοσμιοποίησης, οι μελέτες που έχει κάνει το δικό μας τμήμα δείχνει ότι περίπου το 25% των πλεονασμάτων, των οικονομικών πλεονασμάτων στην ουσία διαρρέει και φτάνει στο επίπεδο του αρχικού μάλλον διαφεύγει του αρχικού παραγωγού, ε, πάει στο εκείνους που κατεργάζονται τα προϊόντα, που επεξεργάζονται τα προϊόντα μετά δηλαδή την παραγωγή του. Ο αρχικός ε, ε, και στην υπόλοιπη αλυσίδα, ο αρχικός παραγωγός δεν χαίρει αυτού του, αυτών των χρημάτων. Γι' αυτό και η Ένωση έχει ε, ε, φτιάξει αυτή την πολιτική ενισχύσεων. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Το πλεόνασμα κανονικά πρέπει να φτάνει στον αρχικό παραγωγό. Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε την κοινή γεωργική πολιτική σε αυτό το πλαίσιο που μόλις σας περιέγραψα στις ε, υποσυνθήκες γενικευμένης παγκοσμιοποίησης οι γεωργοί τείνουν να εστιάζουν την προσοχή στους εμπορικούς, στις εμπορικές πτυχές και όχι σε άλλες πτυχές που δεν εκτιμώνται ιδιαίτερα από την αγορά ή δημιουργούν ε, επιπλέον κόστους. Όπως ας πούμε η μόλις του περιβάλλοντος. Και πάλι η διαρροή του οικονομικού πλεονάσματος ή μάλλον η ανακατανομή των κερδών, ας το πούμε έτσι, χωρίς ε, κοινωνικά ισορροπημένη κοινή γεωρική πολιτική θα ήταν αντιπαραγωγική σε σχέση με τις κοινωνικές μας προσδοκίες. Επιπλέον, το βιομηχανικό πρότυπο καταλήγει σε μια κατάσταση όπου ορισμένες περιφέρειες με λιγότερο πλεονεκτικές συνθήκες βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση ενώ οι τιμές αυξάνονται διαρκώς ιδιαίτερα για τους καταναλωτές. Η ασφάλεια τροφίμων ε, μειώνεται και το βιομηχανικό πρότυπο γεωργίας το πιστεύω πως έχει φτάσει στα ωριά του. τα κριτήρια της ε, μικροοικονομικής λογικής δεν αρκούν για τους καιρού τους οποίους ε, ζούμε. Τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά θέματα είναι εξαιρετικά σημαντικά και στο βιομηχανικό μοντέλο όλα αυτά αγνοούνται. Αυτό λοιπόν που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ατελές. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εγγυηθούμε κάποια θεσμικού τύπου στήριξη ώστε να συμπληρωθεί αυτό, να ολοκληρωθεί αυτό το μοντέλο, ιδιαίτερα σε καιρούς όπου βλέπουμε να λιγοστεύουν οι φυσικοί πόροι. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τα πράγματα από μια νέα προπτική. Εάν θέλετε να δείτε περισσότερα σε σχέση με την σημασία της κοινή γεωργικής πολιτικής, θα πρέπει να λάβετε υπόψη στα εξής, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν ορισμένοι τομεί όπου η κοινή γεωργική πολιτική πραγματικά οθεί την αποδοτικότητα πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον οικονομικό μηχανισμό. Αυτό ισχύει σε τομεί ή σε περιοχέ όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει το ρόλο του δεύτερου πυλώνα σε περιοχέ οπου η μεγάλο βαθμό, όπου δίνεται δηλαδή σημασία περισσότερο στου εξωτερικού παράγοντε και στα δημόσια αγαθά ή, πάση περιπτώσει, να αντιμετωπίζουμε ε, ως δημόσια αγαθά. Η ασφάλεια των τροφίμων, ιδιαίτερα σε φάσεις αυξανόμενης ζήτησης, θα έπρεπε να μεταφράζεται στον ε, αγώνα για ποιότητα και επιπλέον ενημέρωση του καταναλωτή. Το πρόβλημα δηλαδή είναι το να βρεθεί η σωστή ισορροπία και να διατηρηθεί. Από τη μια πλευρά έχουμε οικονομική διαχείριση, οικονομική διακυβέρνηση. Από την άλλη είναι οι πτυχές που σχετίζονται με την κοινωνική και περιβαλλοντική διακυβέρνηση. Αυτά τα τρία θα πρέπει να συνδυαστούν. Γι' αυτό και πιστεύω πω πρόκειται για συστημικό πρόβλημα. Η κοινή γεωργική πολιτική θα έπρεπε να λειτουργήσει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πω οι κοινωνικέ ανάγκε και προσδοκίε διαφέρουν από το ένα κράτο στο άλλο. Η οικονομική κατάσταση διαφέρει. Υπάρχουν δυσαναλογίες τι οποίε όλοι γνωρίζουμε. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ε, ξεπεράσουμε αυτές τις αναλογίες θα πρέπει να αλλάξει ο αλγόριθμος εντός του οποίου λειτουργούμε. Η κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιτυχίες δεν είναι οι ίδιες για όλα τα κρατημέλη. Ωστόσο, ο ρόλος της κοινή γεωργικής πολιτικής θα έπρεπε να είναι η εγγύηση ε, κάποιων καθολικών αρχών, αλλά και η εξασφάλιση πολλών λύσεων, πολλαπλών λύσεων. Και γι' αυτό θα πρέπει να βρεθεί η συμβιβαστική λύση. Και ο αγώνας για τη συμβιβαστική λύση είναι ορατός, αν δούμε και τι υπήρχε στις προηγούμενες δημοσιονομικές προοπτικές, ε, 2007-2013. Για να ολοκληρώσω, ε, εάν συγκρίνουμε να δούμε ποιε είναι οι διαφορέ ανάμεσα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και το υπόλοιπο τη Ευρώπη, σίγουρα το δυναμικό ανάπτυξη όσον αφορά τη γεωργική παραγωγή. Αυτό διαφέρει. Θα σήμαινε δηλαδή ότι η αποδοτικότητα της άμεσης στήριξης θα είναι ψηλότερη από ό,τι στις άλλες χώρες. Αυτή θα είναι μία από τις διαφορές και λιγότερη πίεση όσον αφορά το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει πως έχουμε κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά τη συμβατική βιομηχανική γεωργία, ενώ από την άλλη πλευρά οι μεταφορές, οι αλλαγές μπορεί να είναι πιο ε, δραματικές, πιο, πιο ε, μεγάλες. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ε, τις δράσεις ε, που γίνονται σε περιοχές της υπαίθρου σε μεγάλο βαθμό στις χώρες ε, της Ένωσης στις πρώτες 15. Ενώ στην Πολωνία βλέπουμε ότι έχουμε πολύ νέους γεωργούς, αλλά έλλειψη υποδομής και τεχνολογίας. Αυτό μας περιορίζει φυσικά και οι ανάγκες σε επενδύσεις είναι διαφορετικές. Εάν δούμε μια πιο μακροπρόθεσμη εικόνα του συστήματος, ε, όλα αυτά καθίστανται προφανή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πολλά ενδιαφέροντα ερωτήματα γεννά η ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Θα ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Λετωνίας. για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Γιατί οι ακούσαμε και τον πρώτο πυλώνα. Ο κύριος Τσιμερμάνης λοιπόν έχει το λόγο. Ε, Paldies par iespēju uzstāties šeit, latviešu valodā. ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σα μιλήσω στα λετωνικά, να σα παρουσιάσω την κατάσταση στη Λετωνία. Και ξεκινώ ευχαριστώντας όλους τους βουλευτές οι οποίοι υποστήριξαν τη Λετωνία και έκαναν προτάσεις ε, για τον τρόπο που θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε μέχρι το 2020 τις περιοχές της υπαίθρου να αναπτυχθούν. Θα αναφερθώ λοιπόν στα ζητήματα που θα πρέπει, στα οποία θα πρέπει να δώσουμε το, την περισσότερη προσοχή, δηλαδή το δίλημα μεταξύ επιλογής ε, της γεωργικής ανάπτυξης ή ανάπτυξης πέθρου γενικότερα. Είναι ένα ερώτημα ένα δίλημα που απασχολεί την Ευρώπη, το οποίο έχει να κάνει με τη γενικότερη μεταρρύθμιση, πώς δηλαδή θέλουμε στο μέλλον να παρουσιάζεται η ύπεθρος γεωργία σε όλη την Ευρώπη. Τα τελευταία δέκα χρόνια παρουσιάζεται μια αφέμαξη θα έλεγα κοινωνικο-οικονομική στη Λετωνία με αποχώρηση εγκατάλειψη της υπαίθρου ε, από τον πληθυσμό με ε, πολύ χαμηλή παραγωγικότητα κατάλοιπο της Σοβιετικής περίοδου και συνέπειες πολύ δυσμενής ε, για την λετονική γεωργία μετά την κατάρρευση του σοβιετικού μοντέλου. Βρισκόμαστε λοιπόν ε, τελευταίο τροχός της αμάξης στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. με οικονομικά στοιχεία, γεωργικά οικονομικά στοιχεία, τα οποία ήταν πολύ διαφορετικά αν δεν είχαμε περάσει από αυτό το σοβιετικό καθεστώς. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν αλλάζει. Άλλωστε αυτό εξηγεί και τις ε, διαφορετικές τοποθετήσεις και την ε, ε, συναισθηματική προσέγγιση στη Λετωνία του θέματος της Γεωργίας. Είναι πολλοί λοιπόν οι νέοι οι οποίοι εγκαταλείπουν την Ήπεθρο, πηγαίνουν στις πόλεις και δεν είναι ελκυστική για τους νέους η Γεωργία. Και βλέπουμε εδώ τη μεγάλη απόκληση μεταξύ εσόδων που, καλύτερα που μπορεί κανείς να περιμένει αν εργάζεται στην Ήπεθρο ή αν εργάζεται στην πόλη, στα αστικά κέντρα. Για τη Λετωνία η διαφορά αυτή, η απόκληση αυτή είναι στο 40%. Πολύ σημαντικό ποσοστό, το οποίο δεν ε, μπορεί μόνο να εξηγηθεί με τη διαφορετική ανάπτυξη της υπαίθρου στη χώρα μας, είναι ένα ποσοστό, μια απόκληση που θα πρέπει οπωσδήποτε να συρρυκνωθεί. Μας απασχολεί ιδιαίτερα αυτό και εργαζόμαστε για το στόχο της συρρύκνωση. και στοχεύουμε μέχρι το 2030 να έχουμε μειώσει σημαντικά το ποσοστό αυτό της απόκλησης. Εδώ στη διαφάνεια βλέπετε την, τα ποσοστά των εργαζομένων στη Γεωργία που έχουν πτωτική στάση. Νωρίτερα η συνέντευξη από την ε, Λετωνία παρουσίασε αντίστοιχα στοιχεία. Έχουμε για ένα μικρό κράτος όπως το δικό μας πολύ σημαντική μείωση μέχρι 60% των εργαζομένων στον χώρο της Πέθρου στα τελευταία 8 χρόνια. και κάθε ένας που αποχωρεί από το χώρο της γεωργίας θα απασχοληθεί είτε στις υπηρεσίες είτε στην ε, κατεργασία, κάτι το οποίο δεν μπορούμε βέβαια να λησμονούμε. Τα ποσοστά παραγωγής, τα στοιχεία της παραγωγής δεν παρουσιάζουν τόσο ταχεία ανάπτυξη. ώστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα του περιορισμού της απασχόλησης στη Γεωργία στην Ήπεθρο γενικότερα. Προφανώς προσπαθούμε και εμείς να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα, και τα ποσοστά της απασχόλησης. Είδε μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων στον χώρο της υπαίθρου, 30% περίπου είναι ε, σε προχωρημένη ηλικία, συνταξιούχοι ή στην ηλικία της ταξιοδότησης καλύτερα, χωρίς άλλη πιθανότητα απασχόλησης πέραν της υπαίθρου της γεωργίας. Αυτό οφείλεται και στο μεγάλο αριθμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Λετωνία. Είδε γεωργική δραστηριότητα ε, η οικονομική δραστηριότητα στη Λετωνία ε, συγκεντρώνεται στις μεγάλες, στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ είναι πολύ περιορισμένο το ποσοστό που καλύπτεται από γεωργική γη. 1,4 με 2,2 εκατομμύρια εκτάρια, από τα 2,2 εκατομμύρια εκτάρια που θα μπορούσαν να, να αφιερωθούν στη γεωργική εκμετάλλευση, ε, πολύ χαμηλό ποσοστό δηλαδή, κοντά στο 40%, ε, είναι γεωργικές γεές, ε, που εκμεταλλεύονται, ε, που καλλιεργούνται. Ένα άλλο κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα είναι η γεωργία που πλήθηκε ολόκληρη την Ευρώπη βέβαια, ιδιαίτερα στον χώρο της Πέθρου. Υπάρχουν όμως περιοχές στη Λετωνία που παρουσιάζουν μέχρι και 80% ανεργία. Η τάση πολλές φορές φαίνεται αναπόδραστη γιατί είναι χαμηλότερη ένταση εργασία με τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής στη γεωργία. Και εδώ βλέπετε τα στοιχεία της ενεργείας στη Λετωνία. Με πολύ ανησυχητικές. Εγκατάλειψη της υπαίθρου. που απαιτεί βέβαια την εξέβρεση αποτελεσματικών και καινοτομών μέσων για την ενίσχυση της δραστηριότητας στην Ήπεθρο περιφερειακής ανάπτυξης. Οι μεταναστευτικές τάσεις. 200.000 περίπου Λετωνοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα το 2004 έως 2010 πέραν του φαινομένου της αστιφιλίας. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα μετανάστευσης και ως εκ τούτου έχουμε λιγότερους πολίτες που καταβάλουν φόρο, λιγότερα έσοδα στον εθνικό προϋπολογισμό. Μεγάλο πρόβλημα για τη Λετωνία, ιδιαίτερα καθώς οι νέοι είναι αυτοί που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους, τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και προσπαθούμε να πείσουμε τους νέους να παραμείνουν στην ε, γεωργία, στη χώρα. Αλλά αν δεν έχουν καμία προσφορά, καμία ευκαιρία, ε, στην Ήπεθρο να απασχοληθούν ε, οι νέοι, τότε είτε θα πάνε στο μεγαλωστικό κέντρο είτε θα φύγουν στο εξωτερικό. Βλέπουμε εδώ περιοχές της Ήπεθρου με πολύ αραιό πληθυσμό, ενώ αντίστροφα στα αστικά κέντρα η συγκέντρωση είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε περιοχές στη Λετωνία με πληθυσμό μικρότερο των τριών κατοίκων στο τετραγωνικό χιλιόμετρο, ε, πράγμα το οποίο αποτελεί ρεκόρ για την Ευρώπη, πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Η ανάπτυξη της ε, υπαίθρου ε, κυρίως παρουσιάζεται στις περιοχές γύρω από τα μεγάλα κέντρα, στις περιοχές της υπαίθρου γύρω από τα μεγάλα κέντρα. Υπάρχουν πολλές φορές μάλιστα κάτοικοι της υπαίθρου που παραμένουν στη, στο χωριό τους, αλλά πηγαίνουν καθημερινά στα μεγαλαστικά κέντρα για να δουλέψουν. Ένα άλλο φαινόμενο. Εδώ βλέπετε τις αμοιβέ, μάλλον τις ε, πληρωμές, ε, τις ενισχύσεις κατά έκταση και βλέπετε τις περιοχές της εντατικής γεωργικής εκμετάλλευσης που βέβαια ε, αποκομίζουν την ωφέλη από τις ε, στραματικές ενισχύσεις. Εν τω μεταξύ, ε, τα τελευταία χρόνια, από το 2004 μέχρι τώρα, έχει δεκαπλασιαστεί περίπου η αξία της γης στη Λετωνία. Σε μεγάλο βαθμό αυτό ε, είναι αποτέλεσμα της κέρδοσκοπίας. Αλλά αναμένεται ότι και στο μέλλον θα συνεχιστεί η αύξηση της αξίας των τιμών καλύτερα της γης. Ε, τις εκτάσεις αυτές δεν τις αγοράζουν όμως πάντα γεωργοί. Πρόκειται για χρήμα το οποίο ε, θα έπρεπε να ε, φτάσει στον Γεωργό ως στρωματική ενίσχυση, αλλά εν τέλει δεν φτάνει στις έπαιρες του Γεωργού, αλλά σε εκείνους ε, που έχουν για λόγους κερδοσκοπίας αγοράσει γεωργικές γεές. Για τον Γεωργό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία φυσικά η, ο κοινωνικός περίγυρος, ο κύκλος, ο χώρος, η περιοχή στην οποία ζει κανείς, που μπορεί να βγει το Σαββατοκύριακο, που μπορεί να έχει τον κοινωνικό του κύκλο, που θα έχει τις ευκαιρίες και για την επικοινωνία, όπως είναι πολύ σημαντικό για τους ε, νέους, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε μια περιοχή όπου ε, υπάρχουν τρεις κάτοικοι στο τετραγωνικό χιλιόμετρο, ένας νέος δεν θέλει να κατασταθεί. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Γιατί τα προβλήματα αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Αυτά εν γέννη όσον αφορά τις εξέλιξεις στη Λετωνία. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω αυτές τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Συζήτηση τώρα. Ερωτήσεις. Θα ρωτήσω εγώ την πρώτη ερώτηση στον καθηγητή Τσιρεύσκη. Είπατε, κύριε Τσιδεύσκη, ότι οι συζητήσεις που κάνουμε εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας συχνά καταλήγουν στην ε, εισαγωγή νέων λύσεων. Μάλιστα ότι δημιουργούμε τελικά μια νέα οικονομική πολιτική. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Η γεωργία, η... τα γεωργικά οικονομικά είναι κάτι διαφορετικό από την οικονομία σε άλλους τομείς. Γιατί υπάρχει η γη. Και η γη είναι ο παράγοντας κλειδί για την παραγωγή. Οπότε η γεωργική παραγωγή είναι τελείως διαφορετική από άλλου είδους παραγωγή. Είπατε επίση ότι θα έπρεπε να έχουμε οικουμενικές λύσεις. Καταρχήν, ναι, αλλά βέβαια με κάποια διαφοροποίηση στην πράξη. Το ερώτημα όμως που τίθεται εδώ είναι πώς θα διατυπώσουμε αυτές τις οικονομικές λύσεις που να γίνονται και οικουμενικά αποδεκτές. Και πώς θα καταλήξουμε στη διαφορετική μορφή για να έχουμε λάβει υπόψη μας τις διαφορετικές καταστάσεις της γεωργίας στις διάφορες περιφέρειές μας. Έχω μια ερώτηση βέβαια και για τον δεύτερο μιλητή. Αναφερθήκατε στην πώληση γης ή στη μεταφορά γης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα σε πολλές χώρες μέλη. Το θέμα είναι τελικά ποιος αγοράζει γεωργική γη. Αν είναι το κεφάλαιο, τότε υπάρχει μια στρέβλωση στη γεωργική πολιτική. Γιατί οι μικροί γεωργοί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ένα δυνατό κεφάλαιο. Γι' αυτό και εδώ χρειαζόμαστε καλές λύσεις, ώστε οι γεωργοί να χρησιμοποιούν την γη τους για να παράγουν αγροτικά προϊόντα οι γεωργοί ε, και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν εισόδημα από τη δραστηριότητά τους. Γι' αυτό είναι δύσκολο εδώ να έχουμε λύσεις. Και ένα άλλο πρόβλημα είναι πιο αραιοκατοικημένες περιοχές. Βλέπω ότι ο κύριος Γιάρ επίση θέλει να ρωτήσει κάτι. Είσαστε έτοιμος για την ερώτησή σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Α, έτσι κι αλλιώ ε, είσαστε πάντα απαραίτητο εδώ στην Επιτροπή μας. Ε? Σας ακούμε. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω ε, το θέμα της οικονομικής ε, πολιτικής στον χώρο τη υπαίθρου είναι πολύ περίπλοκο και δύσκολο και πρέπει να συζητηθούν πολλά θέματα, να δοθούν ευκαιρίε και λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να είναι ποτέ γενικές δεν μπορεί να ισχύουν για ολόκληρη μια περιφέρεια χωρίς διαφοροποίηση. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν. Ήταν σχετική με την κερδοσκοπία στη γη. Όταν σημαίνει αυτό, η λειτουργία του υπαίθρου ως ευκαιρία για την δημιουργία θέσεων εργασίας ε, χάνεται. Πρέπει λοιπόν νομίζω να μεριμνήσουμε εμεί από την ευρωπαϊκή πλευρά οι πληρωμέ ε, του πρώτου πυλώνα να μην πηγαίνουν στον γεωκτήμονα, αλλά στον εργάτη της γης, στον γεωργό. Αυτό πιστεύετε ότι θα αρκούσε ή θεωρείτε ότι χρειάζονται παραπάνω μέτρα. Και δεύτερο ερώτημα για την, για την οικονομική πολιτική. Η στρατηγική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής μας με τον πρώτο πυλώνα και την ανάπτυξη πέθρου ε, συνοδευόταν και από το Ταμείο Συνοχής το οποίο είναι διαρθρωμένο έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν το δικαίωμα της συνδιαμόρφωσης των πολιτικών για τις περιφέρειες, να μην επιβάλλονται δηλαδή αποφάσεις από τις Βρυξέλλες για το τι συγκεκριμένα χρειάζεται μία περιοχή. για να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση ή θέσεις εργασίας. Ερωτώ λοιπόν, βλέπετε να υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί και έχετε δει μηνύματα ότι αρκούν αυτά που κάνουν οι Βρυξέλλες ή έχετε και άλλες συστάσεις, γιατί εγώ νομίζω ότι ε, δεν ε, δει μόνο χρημάτων. Υπάρχουν ε, άλλες λύσεις στρατηγικές και σχέδια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Βλάτφερντ, αν δεν απαιτώ με θέλει το λόγο. Αν δεν θέλει κανείς άλλος το λόγο. Τότε παρακαλώ να λάβουν ε, το μικρόφωνο οι δικοί μας για να απαντήσουν οι πυρογνώμονες. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω γιατί κάποιες από τις ερωτήσεις σας απευθύνονταν σε μένα προσωπικά. Λοιπόν, Πρόεδρε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η κατεύθυνση παίζει καθοριστικό ρόλο. Η κοινή γεωργική πολιτική διαμορφώνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πολύ συχνά πρόκειται για λύσεις ad hoc. Δηλαδή προκύπτει ένα πρόβλημα, άρα πρέπει να βρούμε μια λύση. Και συνεχίζουμε. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι διαμορφώνουμε μια πραγματικά διαφορετική αγροτική οικονομία. Εγώ αναφέρθηκα σε νέα αγροτική οικονομία ενώντας ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται θα πρέπει να μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε κάτι το οποίο δεν είναι ορατό με διαγυμνού οφθαλμού. Μιλάμε για έσοδα που έχουν να κάνουν με την ταξινόμηση της γης. Αν η ζώνη στην οποία βρίσκεται η γη αυτή θεωρείται απομακρυσμένη, μειονεκτική. Τα πράγματα αλλάζουν. Η κατάσταση σήμερα είναι τέτοια όπου το 1 τρίτο των αποβλήτων δεν απορροφείται τελικά από τη φύση. Γιατί δεν έχει πια την ικανότητα αυτή η γη να απορροφήσει τόσο μεγάλες ποσότητες αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πήρε μια καλή απόφαση στο δεύτερο πυλώνα λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή διάσταση το περιβάλλον. Και εδώ έχουμε ηγετικό ρόλο, παγκοσμίω. Οι Αμερικανοί είναι πίσω από μας και η Ασία ακόμα πιο πίσω. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια καλή κατεύθυνση που έχουμε πάρει. Και δεν είναι επειδή θέλουμε να πάμε τόσο μπροστά, αλλά επειδή οι ανάγκες μας ήταν τέτοιες που απαιτούσαν κάποια απάντηση μια δεδομένη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τη νέα αγροτική οικονομία και να εισαγάγουμε στην οικονομική διάσταση όλους αυτούς τους παράγοντες που δεν έχουν ληφθεί υπόψη μέχρι τώρα και που είναι η αξία της γης γιατί από εκεί απορρέει αξία που όμως μέχρι τώρα την κερδίζουν οι... την κερδίζουν άλλοι και όχι εμείς. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι είναι δύσκολο. Μπορεί να είναι δύσκολο και για τον Γιώργο. Γιατί αν μιλούμε για την εγγενή αξία της γης, πρέπει να συζητήσουμε και την εγγενή αξία τον υδάτωνε, παραδείγματι, και να πείσουμε τους γεωργούς ότι τον κάθε γεωργό ότι το νερό στο πηγάδι του δεν είναι μόνο δικό του, ότι είναι ένα κοινό αγαθό, ένα δημόσιο αγαθό και με κάποιο τρόπο πρέπει να υπολογιστεί η αξία του. Ή όταν ένας γεωργός δεν τηρεί τους όρους του greening, της πράσινης ε, γεωργίας. Πάλι θα πρέπει να υπάρχουν συνέπειες. Εσείς μιλήσετε για παγκόσμιες ε, οι οικουμενικές λύσεις, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, μόνο οι αρχές μπορούν να είναι οικουμενικές. Τα προγράμματα, τα σχέδια, τα συστήματα θα είναι εθνικά. Υπάρχει το οικουμενικό βέβαια σύστημα της ε, προσφοράς και της ζήτησης που φέρνει πάντα αποτελέσματα, αλλά θα πρέπει και να προσδιορίσουμε το κόστος και το εισόδημα κόστος και έσοδο και το πώς θα υπολογιστούν αυτά στην πράξη. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πρακτικό ζήτημα, το οποίο ανά περιοχή θα πρέπει να ε, αξιολογηθεί. και να δοθεί μια σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από την ε, κατεύθυνση που έχει επιλεγεί. Ε, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε, να ενσωματώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τον επόμενο μιλητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. το πρόβλημα της ε, αγοράς ε, γης ε, από μη γεωργούς είναι ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό. Έχουμε να κάνουμε μεγάλους επενδυτές που αγοράζουν γη. Έχουμε να κάνουμε ένα φαινόμενο δεδομένο στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, της Βαλτικής ιδιαίτερως, και θα πρέπει να σκεφτούμε το πρόβλημα διαφορετικά γιατί έχουμε εξαρτήσει για, τη, για τα έσοδα, για τα εισοδήματά τους αυτούς τους γεωργούς από τις ε, άμεσες ενισχύσεις και για την επιβίωσή τους αλλά από την άλλη ε, θα μπορούσαν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Και δεν μπορούν εκμεταλλεύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν πιο αποτελεσματικούς τρόπους παραγωγής να ε, πάρουν εκτάσεις ε, γεωργικές γιατί κάποιοι δεν είναι τυθμένοι να τις πουλήσουν. Αρκούν λοιπόν αυτά που κάνουμε. Ένα πρόβλημα ότι αισθάνεται ο Γιώργος ότι δεν έχει ε, ισότιμη αντιμετώπιση. Χρειάζονται λοιπόν περισσότερες επενδύσεις στη Γεωργία. Οι μεγάλες υποδομές και οι επενδύσεις στις μεγάλες υποδομές προχωρούν περισσότερο στα αστικά κέντρα και πολύ λιγότερο στην Ήπεθρο, παρότι οι μεγάλες ανάγκες εντοπίζονται στην Ήπεθρο, αλλά επειδή είναι πολύ πιο ακριβά, ε, ακριβές οι επενδύσεις και αραιός ο πληθυσμός δεν γίνονται οι επενδύσεις στην Ήπεθρο. Υπάρχουν περιπτώσεις μάλιστα όπου ο άξονες ούτε καν επισκευάζονται, ούτε καν συντηρούνται και έτσι επιδεινώνεται και επιταχύνεται ακόμη περισσότερο αυτή η τάση των πολιτών να καταλήγουν την Ήπεθρο. μία ευκαιρία, μία δυνατότητα την οποία δεν έχουμε αξιοποιήσει παρκώς από την εμπειρία μας από τη σχεδιασμένη σοβιετική οικονομία. Θέλω ότι μπορούμε να διαγνώσουμε ένα θετικό, ένα δυναμικό, ότι έχουμε δυναμικό ανάπτυξης ε, κατά 80-90% περισσότερο από ότι τώρα. Δεν μπορούσαμε ακόμη το δηλαδή να αναπτυχθούμε και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλήρως αυτό το δυναμικό ανάπτυξης. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται να το αναπτύξουν αυτό το δυναμικό, αλλά χρειάζεται, χρειάζεται γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη και για γεωργική οικονομία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνεδρίαση, εκτός βέβαια αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο για κάτι, κυρία Καλιέτε. Δεν ε, μιλήσατε καθόλου σήμερα. Στην επόμενη. Δεν βλέπω κανένα να θέλει να πάρει το λόγο. Θα τελειώσουμε εδώ λοιπόν τη σημερινή μας ακρόαση. Ο τίτλος της σημερινής ακρόασης ήταν να συζητήσουμε τις εμπειρίες των ε, νέων χωρών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ξεκινώντας από το 2004 ή ακόμα και πριν την ένταξη. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τι σήμαινε η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές τις χώρες. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι σήμαινε πως μπαίνανε σε ένα εντελώς νέο σύστημα οικονομικό, πολιτικό, δημοκρατικό, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σίγουρα οι επιπτώσεις στην Ήπεθρο ήταν τεράστιες δεδομένου ότι η Ήπεθρος συχνά βρισκόταν πολύ πιο πίσω όσον αφορά την ανάπτυξη. Και για να απαντήσω και στην ερώτηση της κυρίας Μαγκίνες, ναι, το επίπεδο ζωής στην Ήπεθρο έχει αυξηθεί πολύ. Και αυτό γιατί έχουν εφαρμοστεί αλλαγές που δεν υπάρχει περίπτωση να αντιστραφούν τώρα. Σίγουρα όμως υπάρχουν και διαφορές. Υπάρχει πιο βιομηχανική γεωργία, υπάρχει πιο οικολογική γεωργία. Είχαμε μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και το μέγεθος της παραγωγής ήταν πολύ μεγάλο. Μετά άλλαξε η κατάσταση και τώρα υπάρχουν διαφορές στα μεγέθη. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι μία λύση ταιριάζει σε όλους. Πάντως η ανταγωνιστικότητα είναι ένα πολύ βασικό κριτήριο όταν μιλάμε για οργική πολιτική. Ίσως δεν ασχοληθήκαμε αρκετά με την ε, διατροφική ασφάλεια. το θέμα αυτό επίσης έχει βελτιωθεί μετά την ε, ένταξη και αυτό γιατί έχουμε ε, μεγαλύτερες αγορές, ε, μεγαλύτερη πρόσβαση σε προϊόντα καλής ποιότητας και έπειτα υπάρχει και λειτουργία της σημερινής αγοράς που αναφερθήκαμε σε αυτήν. Οπότε για το μέλλον της ΚΑΠ Ξέρω ότι είναι κάτι που συζητιέται στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου, πάντως το συμπέρασμά μου εμένα είναι ότι όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα εμπλουτίζουν και τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν ε, το πρόβλημα ή τη λύση αν είναι η λύση, τότε πρέπει να φροντίσουμε να εφαρμοστεί αυτή η λύση. Ποιο όμως θα πληρώσει τελικά το λογαριασμό γι' αυτό. Συχνά έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε ότι οι μικρές γεωργικέ εκμεταλλεύσεις μπορούν να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο όπως και οι μεγάλες. Δεν ισχύει όμως αυτό. Μια μικρή γεωργική εκμετάλλευση δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αντιγράψει την απόδοση και την σοδιά μιας μεγάλης. Χρειάζεται έτσι κι αλλιώς διαφορετικό μοντέλο. Έπειτα, η... ο χώρος παραγωγής και ο χώρος όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση στην παραγωγή καταναλωτές. Η διαφορά αυτή. Πώς μπορούμε να καταφέρουμε να βάλουμε, πώς να σας το πω, το κουβέρ του καταναλωτή δίπλα στον αγρό όπου παράγεται το αγροτικό προϊόν. Η κοινή γεωργική πολιτική εδώ θα έπρεπε να βοηθήσει. Το θέμα της υποδομής τέλος έχει μεγάλη σημασία γιατί αν δεν έχουμε την κατάλληλη υποδομή δεν μπορούμε να λύσουμε και τα προβλήματα τα οποία σήμερα είναι πολύ σημαντικά για τον αγροτικό χώρο. Εδώ ολοκληρώνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να ξέρετε ότι είναι έτσι κι πολύ δύσκολη Δευτέρα κάθε εβδομάδα γιατί μερικοί δεν προλαβαίνουν να έρθουν εδώ στην ώρα τους, άλλοι από εμά ε, ε, είχαμε, λείπαμε από την Παρασκευή και κάποιοι δεν έχουν γυρίσει ακόμα. Πάντως με τους εμπειρογνώμονες πιστεύω ότι καταφέραμε να συζητήσουμε καλά, έγιναν ερωτήσεις και αυτοί που δεν ήταν εδώ θα ενημερωθούν για τα συμπεράσματα της συζήτησής μας. 29 Μαΐου είναι η επόμενη συνεδρίασή μας και 30 Μαΐου. Ξεκινάμε την 5η δηλαδή στις 3. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, λίγη εδώ η σημερινή συνεδρίαση. Καλό βράδυ και άλλη μια φορά ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες. Οι παρουσιάσεις σας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες να ξέρετε και ελπίζω ότι η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί και στην Κρακοβία, στην ε, στο συνέδριο που θα έχουμε εκεί τον Ιούλιο. Θα είναι η τρίτη διάσκεψη αφιερωμένη σε αυτό ακριβώς το θέμα. Ελπίζω να βρεθούμε με τους εμπειρογνώμονές μας στην Πολωνία τότε λοιπόν. Σας ευχαριστώ.